Colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Ας ξεκινήσουμε την ε, πρωινή συνεδρία με την ε, έκθεση της συνάντησης των συντονιστών. Καταρχάς, σε σχέση με την ονομασία των, ε, με τον ορισμό των εισηγητών, οι συντονιστές αποφάσισαν ότι μόνο σε μία εκ των εκθέσεων που είναι συμφωνία για τις ελαμπορικές υπηρεσίες μεταξύ Ευρω... Ευρωπαϊκής Ένωσης και της, ε, και της ε, Δημοκρατίας του Πράσινου Ακροτηρίου θα πρέπει να γίνει σχετική έκθεση. Η άλλη, σε ό,τι αφορά τη χαρτογράφηση ενός περιβάλλοντος κοινή ανταλλαγή στοιχείων για το κοινοτικό περιβάλλον ναυτιλίας δεν θα λυθεί η δράση. Ευχαριστούμε την Επιτροπή που προσπάθησε να δώσει τα μεγαλύτερα και τα πιο μακριά ονόματα σχετικών ανακοινώσεων και εκθέσεων που μπορεί να σκεφτεί σε σχέση με τα έγγραφα για την ανταλλαγή πληροφοριών και αγρομοδοτήσεων, ανακοίνωση του προγράμματος 11 συντονιστές αποφάσισαν να λάβουν σχετική δράση και λόγος είναι ότι οι πολιτικές ομάδες σίγουρα θέλουν να συσφέρουν ισχυρά στο πρόγραμμα εργασίας του 2011, αν και τονίστηκε από τους συντονιστές ότι τα μέλη στις διάφορες πολιτικές ομάδες θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι μεταφορές και ο τουρισμός να μην παραβλεφθούν. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν επαναφέρουμε και επαφιόμαστε σε εσά ω καλούς συμπροβουλευτές να πολεμήσετε το συγκεκριμένο ζήτημα όταν οι πολιτικές ομάδες συζητήσουν τη θεματική αυτή. Σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση της αναθεώρησης του κοινωτικού προπολογισμού, αναβλήθηκε η απόφαση γιατί ακόμα δεν αποφασίστηκε την Επιτροπή Προπολογισμού τι μορφή θα λάβει στην Επιτροπή. Όπως ξέρετε υπάρχουν εξελίξεις διαπραγματεύσεις στον ε, ε ενισχύ προϋπολογισμό. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει λοιπόν. Η αποφάση λοιπόν θα αναβληθεί ως ότου ε, δούμε ακριβώ τι θα κάνουν οι συνάδελφοι της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Σε ό,τι αφορά τη σχέση με τα Εθνικά Κοινοβούλια, οι συντονιστές ακολούθησαν την πρόταση του Προέδρου. Οι ακόλουθοι ε, φάκελοι η πρόσβαση στη δρομική, αγο... στη δρομική αγορά, η ασφάλεια των αέριων μεταφορών και η συνεργασία μεταξύ των Αθηνικών Κοινοβουλίων μπορούν να γίνουν μέσω των εισηγητών των Επιτροπών Μεταφορών που θα είναι υπεύθυνοι για του φακέλου αυτού, οπότε οι εισηγητέ θα μπορούν στη συνέχεια να ενημερώσουν του συντονιστέ. Και οι φάκελοι αυτοί είναι τμήμα του, είναι ανεπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος εργασίας 2011. Ε, Σε ό,τι αφορά τώρα την επιτροπολογία, πληροφορώ τις ε, συντονιστές ε, της, ε, του προσχέδιου απόφαση Επιτροπής σε ό,τι αφορά τους νέους κανόνες για την παρακολούθηση και την ασφάλεια του εναέριου αέρα του, του αναέριου χώρου. Το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα παρακολούθηση για ένα μήνα. Ο εισηγητή, ο κ. Βασπάλ, θα προσκληθεί να εξετάσει το ζήτημα αυτό στην έκθεσή του στα θέματα ασφάλεια αέριων μεταφορών, στην αρχική έκθεση πρωτοβουλία την οποία αναλάβει και την οποία συντάσσουμε. Τώρα στα διάφορα, ο πρόεδρος θα είναι εισηγητής για γνωμοδότηση στην Επιτροπή. Η εργασία αυτή είναι ήδη εξελίξη και θα προσπαθήσουμε να την ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν. Αν έχει κανείς κάποια ερώτηση, αυτά σε ό,τι αφορά την εργασία των συντονιστών. Αν όχι, συμφωνούμε ότι ούτως έχει. Θεωρείται ότι το έχουμε κρίνει. Ευχαριστώ. Επόμενο θέμα. Όλοι αναζητούμε τις ε, κάρτες μας για την ψηφοφορία. Θα ξεκινήσουμε με την, ε, με υποχρεωτική δοκιμαστική ψηφοφορία. Εάν όλοι έτοιμοι λοιπόν με τις κάρτες ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχουν ψηφίσει όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Ωραία. Εντάξει, είναι πάντες ο κ. Κομουτσάκος. Μα όταν φτάνει στη σοφορία μας το λέτε. So, first vote is the... Έκθεση Σίμψον περιστατιστικών στον τουρισμό. Ξεκινώ με την τροπολογία 21. Θα το έλεγα. 21, 23 και 24 έχουν αποσυρθεί. Οπότε, επόμενη τροπολογία. Τροπολογίες 4, 6, 11, 12, 17. Όλες μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Επόμενη τροπολογία 22. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 3 του συγητή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7, 11 και 12 σελίδιν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25, κυρία Ντιουράν, κύριος Κράμερ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 του κυρίου Κόζα με προφορική τροπολογία που θα πρέπει να έχει ψηφιστεί από τον κύριο Φιντάντσα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 Υπέρ, εδώ πέρα γίνεται έλεγχος ασφαλείας για το ΕΛΚ που θα ακολουθήσει, εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχή. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στα παρατήματα. Πετροπολογία 27 του κυρίου Κόζα υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγξουμε την τροπολογία του κυρίου Κόζα. Τροπολογία 27. η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα ψηφοφορία. 22 υπέρ. Συγγνώμη, 34. Ψήφισαν 22 υπέρ, 12 κατά. Υπερψηφίστηκε. 28 Ντυράν και Κρέιμερ υπέρ Συγγνώμη, 28 και 30 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά αποχές θα το ελέγξουμε. Τροπολογία 32 του κυρίου Φιντάντσα. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψήφισαν όλοι. Πέρα 20 υπέρ, 15 κατά. Νομίζω αλληλοαποκλειστήκατε. Ωραία, εγκρίνεται. Τώρα, στην αιτιολογική έκθεση Επαριθμό 2 με προφορική τροπολογία λόγο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1 υπέρ. Θέλετε να αλλάξουμε. Ο επικεφαλής του ΕΛΚ φαίνεται ότι διαφωνεί με την ομάδα του. Λοιπόν, ελέγχουμε. Τροπολογία 18. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογία 18. Ψήφισαν όλοι. Πέρα 10 υπέρ, 27 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19. Κυριατικά. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 κυριατικά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τροπολογία 2 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα, τη χτίση ψηφοφορία η όλη νομοθετική πρόταση κατόπιν τροπολογιών, η ηλεκτρονική του ψηφοφορία. Έναρξη. Κύριε αυτή την κάρτα έτσι. Είναι ενδιαφέρον, γιατί αμέσως μόλι πήρατε την κάρτα σας, έχει, υπάρχει μια πρόσθετη ψήφο στο ΕΛΚ. Πολύ ενδιαφέρον. Μπορεί κάποιο από το ΕΛΚ, παρακαλώ πολύ, να αποσυρθεί. Πολύ ωραία. τη ψηφορία. Δεν νομίζω ότι έκανε και πολύ μεγάλη διαφορά. 37 ψήφισαν, 37 υπέρ, καμία κατά, καμία αποχή. Οπότε το νομοθετικό, το νομοθετικό ψήφισμα, έναξη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορία. 34 ψήφισαν, 34 υπέρ, κανείς κανά, καμία αποχή, επομένως εγκρίνεται ομοφόνος. Και τώρα, μιας και έχουμε αυτή την υιοθέτηση την ε, σαρωτική από την Επιτροπή. Ελπίζω η Επιτροπή να μου δώσει μια εντολή επί τη βάση της μη ψηφοφορία να πάω να πραγματευτώ με το Συμβούλιο. Είστε ευτυχείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα το Συμβούλιο θα προσβλέπει με πολύ μεγάλη ανακούφιση τη διαπραγμάτευση αυτή. Και τώρα, επόμενη ψηφοφορία, η έκθεση του κυρίου Κράμαρ σχέδιο έκθεσης ε, για την πολιτική ανταγωνισμού του 2009 στο πεδίο των μεταφορών. Καταρχάς, βρισκόμαστε στην παράγραφο 1. Συμβαστική πρόταση Α. Ποιοι είναι υπέρ. Παριέσαι τρελά, θες. Εγκρίνεται. Ερχόμαστε στην τροπολογία 4. Κύριε Ζέλη, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Those against. Abstention. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οκτώ υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίπτεται αλλά να ελέγξουμε λίγο παρακαλώ πολύ τροπολογία 8 Ένα πληροφορίας. ψήφισαν όλοι Πρωτού την κλείσω, το ΕΛΚ πάλι έχει μία ψήφο παραπάνω. Εντάξει. Πέρας ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 23 κατά. Καταπίπτει. Απορρίπτεται. 9. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εάν διαγράφεται η 10 Είσαι εδώ. Πολύ ωραία. 10. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το ελέγξω. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θέλω να το ελέγξω. 13. Wortman Call. Έναξη πληροφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα πληροφορία. 27 υπέρ, 11 κατά, σαφέστα εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 15 και 16. καταπίπτει γιατί 14 εγκρίθηκε, έχετε δίκιο. Και η 17 λοιπόν το ίδιο, οπότε περνάμε στο 18. Ο εισηγητής, προφορική τροπολογία. Θέλουμε να, να κρατήσουμε την ξεχωριστή ψηφοφορία και αντιτιθέμεθα στην προφορική τροπολογία. Καταρχά να το θέσω. Υπάρχει προφορική τροπολογία του κυρίου Ρικέ εκ μέρου του ΕΛΚ. Υπάρχουν αντιρρήσει προ την προφορική τροπολογία. Εσεί, ο εισηγητή. Ως εκ τούτου δεν μπορώ να την θέσω σε ψηφοφορία, εφόσον υπάρχει αντίρρηση σχετικά. Και ζητήσατε ξεχωριστή ψηφοφορία. Περί πού ακριβώς. Σε ποιο στο 18. Σε ποιο σημείο στο 18. Κύριε Στάξη. Υπήρχε ένα αρχικό ερώτημα που είχε τεθεί από το ΕΛΚΕ, ζήτημα να γίνει χωριστή ψηφοφορία ή να ξεχωριστούν ψηφοριστά πάνω στις, ε, για τις λέξεις που ήταν εντός εισαγωγικών. Έχει κανείς αντίρρηση σε αυτή τη ξεχωριστή ψηφοφορία? Εάν όχι, παίρνω την διατύπωση χωρίς την ε, φράση εντός εισαγωγικών. Εντάξει, ποιοι είναι υπέρ της τροπολογίας 18 χωρίς τις, τα εντός αγωγικών. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, με τη διατύπωση αγωγικά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η φράση εντός αγωγικών. 22 κύριε Ζήλαντ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 και 22. Το 22 δεν ακριθεί, οπότε δεν καταπίπτει. 21 και 22. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 απο, αποσύρεται 24 ξεχωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα μέχρι τις βιομηχανίες δεύτερο όπως το εμπόριο πρώτο κομμάτι ποιο είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο κομμάτι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προπολογία 28 του κ. Ζήλα, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 26 και 27 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Abstentions. Να αλλάξουμε το 30, Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. many again. Το ΕΛΚ. Πάλι μία ψήφο παραπάνω. Πέρας ψηφοφορίας. 21 υπέρ, 14 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 31, ως προσθήκη. Υπέρ, κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 31 παρακαλώ. Της ως προσθήκη. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσαν όλοι. πέρα ψηφοφορίας. 13 υπέρ 37 κατά απορρίφθηκε. 32 αποσύρθηκε. 33. Αντί του 32 χωριστή ψηφοφορία για την παράγραφο 8 σε δύο τμήματα. Το πρώτο μέρος καλεί την Επιτροπή για να μπορεί να εφαρμοστεί και το δεύτερο μέρος θα καταπίσει αν δεν εγκριθεί το πρώτο. Ψηφίζουμε λοιπόν για την παράγραφο 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 33. Τικάου. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 34. Στέρξ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 35. Δερικέ, υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 36. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 37. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός Β. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Πάμε στην 41, στέρξ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 43, και 40, και 40 καταπίπτουν, 42 τικάου υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 45 τικάο υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός γάμα υπέρ κατά αποχές θα ελέγξω με το συμβιβασμό γάμα αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 19 κατά, κατά πίπτη. Τελική ψηφοφορία. Συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε ακόμα και δύο άλλες τροπολογίες. 23 τικάο υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 44 στέρξ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Αυτό ήταν χρήσιμο συνάδελφοι. Περνάμε λοιπόν στην τελική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. everybody voted. Ψήφισαν όλοι. Πέρα ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 3 κατά, 7 αποχές, εγκρίθηκε συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ευχαριστούμε συνάδελφοι. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη Is the Είναι αεροπορική ασφάλεια με ιδιαίτερη έμφαση στους σαρωτές προτού καλέσω τον κύριο Ντεγκράντες Πασκουάλ θα περιμένω να φύγουν όλοι όσο γίνεται πιο ήσυχα όσοι αποχωρούν παρακαλούνται να φύγουν αμέσως και οποιασδήποτε συζητήσεις που θέλουν επιγόντως να κάνουν, να τις κάνουν έξω παρακαλώ, έξω από την αίθουσα. Okay. Okay. Right. So, very topical at the moment is aviation security. So. Λοιπόν, ασφάλεια, ασφάλεια, αεροπορική ασφάλεια, <clears throat> εισηγητής Λουίς Γκράντες Πασκουάλ. Λουίς, έχει το, έχεις το λόγο. Muchas gracias, señor presidente. Queridos colegas, είναι ένα σημαντικό και επίκαιρο θέμα. Γι' αυτό σας παρακαλώ να δείξετε επίοικια. ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το θέμα αυτό, όπως το, το ε, επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η οικονομική κρίση οπωσδήποτε μας έχει κάνει όλους πιο ευάλωτες και η τρομοκρατία είναι ένα φαινόμενο που έχει πλήξει πολλές χώρες. Η τρομοκρατία είναι μια σοβαρή απειλή ανεξάρτητα από τα αίτια του. Μια απειλή που αντιμετωπίζουμε όλοι. Σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε πράξη τρομοκρατίας. Γι' αυτό οι αρμόδιες αρχές πρέπει να υιοθετήσουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν την ε, προστασία των πολιτών τους. Συχνά, τα μέτρα στον τομέα της ασφάλειας σημαίνουν μείωση των ατομικών ελευθεριών, περιορισμό των ατομικών ελευθεριών που ενοχλεί, ενοχλεί τους πολίτες. Κατά την άποψη της, του εισηγητή, οι πολίτες όμως θα ήταν έτοιμοι, θα ήταν πρόθυμοι να στερηθούν μέρος της ελευθερίας τους για να προστατεύσουν, για να προστατευτούν οι ίδιοι. Τα δημοκρατικά θεσμικά όργανα, ωστόσο, απαιτούν, απαιτούν να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και προστασία για τους πολίτες τους, χωρίς να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Όταν υπέβαλε την πρότασή της το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζήτησε, ήταν αυτό μια αντίδραση σε αυτά που είχαν συμβεί στον κόσμο. Κατά την άποψή μου, η πρόταση ήταν τελείως αυτοσχέδια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, το υπογράμμισε αυτό Βεβαίω, η πρόταση της Επιτροπής στηριζόταν στην καλή πίστη, ε, είχε γίνει με καλόπιστο πνεύμα, αλλά, αλλά ε, κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έπρεπε να περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένα στοιχεία για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. Και ποια ήταν η αντίδραση των κρατών μελών. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες για την αεροπορική ασφάλεια οδήγησε σε διαφορετικές αντιδράσεις στα διάφορα κράτη-μέλη η χρήση των σαρωτών με διαφορε... που στηρίζονται σε διαφορετική τεχνολογία δημιουργεί κάποια προβλήματα και υπάρχει συχνά η ανάγκη για τους ε, ταξιδιώτες να περνάνε από παραπάνω από έναν ε, σαρωτή ε, στη διάρκεια του ταξιδιού τους. Γι' αυτό και και υπάρχει δυνατότητα για τους πολίτες, για τους πολίτες να αντιδράνε σε αυτή τη διαδικασία. Το Κοινοβούλιο έχει θεσπίσει ψηφίσματα για τις επιπτώσεις ε, της χρήσης των σαρωτών, αυτών των σαρωτών και προέβη σε μια εκτεταμένη ανάλυση του θέματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνόψισε ε, και σχολίασε τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αξιολόγηση για την υγεία, με αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε στα συμπεράσματά της ένα δύο σημαντικά σημεία την ανάγκη εφαρμογής των κανόνων με ομοιόμορφο τρόπο ώστε να υπάρχει ισότητα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και να προστατεύεται η υγεία των, με αποτελεσματικό τρόπο των πολιτών, των ταξιδιωτών σε όλα τα αεροδρόμια. Επίσης, εξέτασε τη δυνατότητα εφαρμογής ελάχιστων κανόνων σε ό,τι αφορά τον, τις, τεχνικές, τις τεχνικές προδιαγραφές για αυτά τα μηχανήματα ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος που χαρακτηρίζει τη χρήση αυτών των σαρωτών για την υγεία των ανθρώπων. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια επικοινωνία, ένας διάλογος μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων για να προχωρήσει αυτή, αυτό το θέμα. Ο εισηγητής πιστεύει ότι πρέπει να προβούμε σε μια θετική αξιολόγηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής, διότι η Επιτροπή αναφέρεται στις αμφιβολίες που είχε εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που περιέχονται στο ψήφισμα της 20 Οκτωβρίου 2008 μετά την εφαρμογή ευρωπαϊκών κανόνων για τους σαρωτές υπάρχει τώρα μια νέα γενιά μηχανημάτων που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών. Αυτοί οι σαρωτές προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην αποτελεσματικότητα των ελέγχων ασφαλείας στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια εισαρωτές, τα κράτη-μέλη που θα που θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν αυτούς τους αρωτές, θα πρέπει να τηρούν απόλυτα τους κανόνες που θα ε, θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, επειδή το, το δικαίωμα στην υγεία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, χρειάζεται να, να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες, τεχνολογίες οι οποίες εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή προστασία του ανθρώπινου σώματος. Να αποφεύγονται οι ακτίνες Χ για να μην ε, επιβαρύνονται τα, οι ταξιδιώτες με πρόσθετη ακτινοβολία και να απαγορεύεται η αποθήκευση, αποθήκευση των δεδομένων που λαμβάνονται από τους αρωτές. Στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας, στην κανονισμό 300 του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί στις αναγκαίες αλλαγές. Αυτά που συνέβησαν στην Ιεμένη δείχνουν ακριβώς ποια είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε. οι αεροπαρικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων είναι ο πιο αποτελεσματικός είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για τους τρομοκράτες να σπείρουν παντού το φόβο. Είναι απαράδεκτο από ηθική άποψη τα, θεσμικά, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μην είναι σε θέση να αντιδράσουν σε αυτές τις καταστάσεις πρέπει να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά θα ήταν κατά την άποψή μου ανεύθυνο να παραμείνουμε παθητικοί, αδρανείς, χωρίς να αντιδράμε με αποφασιστικότητα και με αποτελεσματικότητα στις ενέργειες, στις παράδεκτες αυτές πράξεις των τρομοκρατών. Οπωσδήποτε τα μέτρα και τα συστήματα ασφαλεία μας δεν είναι τέλεια, αλλά πρέπει να λάβουμε αποφάσεις. Πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε, να προοδεύσουμε στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας των επιβατών σε θέματα ασφάλειας. Δεν είναι ανάγκη, δεν είναι απαραίτητο όλα να δημοσιοποιούνται. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικά και να μην αποκαλύπτονται, διότι δεν πρέπει να δίνουμε ε, στους εχθρούς της δημοκρατίας ε, πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν, θα χρησιμοποιηθούν εναντίον μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εξηγήσουμε σε όλους ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχουμε όλα, ό,τι, όλα αυτά που χρειάζονται για να αντιδράσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να ε, επιβάλλουμε μια συγκεκριμένη θέση μετά από δικές σας υποδείξεις. Έχουμε μόνιμη, μόνιμη επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε έρθει σε επαφή, έχω έρθει σε επαφή και με τους σκιώδεις δήμερός. Και όταν συμφωνήσουμε, κάποια μέρα θα μπορέσουμε, όταν μπορέσουμε θα ορίσουμε τις μεγάλες κατευθυντήριες γραμμές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα τελευταία γεγονότα που γνωρίσαμε ως προς τη μεταφορά του ταχυδρομείου, ε, φορτίου ή επιβατών. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την Επίτροπη στα πλαίσια της Επιτροπής Μεταφορών κατά πόσο μπορούμε να διευρύνουμε αυτή την ε, έκθεση και θα ήθελα μία ανακοίνηση από την Επιτροπή. Δεν θα πρέπει να περιοριστούμε σε θέματα ασφάλειας, θα πρέπει να ασχοληθούμε ευρύτερα με τους κινδύνους της αεροπλοείας. Γι' αυτό θα πρέπει να ακούσουμε τους πάντες, να, ακολουθούμε, να παρακολουθούμε την επικαιρότητα και να μπορέσουμε με ευθύνη να εγκρίνουμε μία έκθεση μέσα στα πλαίσια μιας διαθεσμικής συνεργασίας, έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και να τηρήσουμε, να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα βεβαίως, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστούμε κύριε Ντεγκράντες Πασκουάλ για να σας απαντήσω. Όπως σας είπα, οι συντονιστές σας ζήτησα να επεκταθείτε έτσι ώστε να δείτε και το θέμα του κάργο. Και βεβαίως λόγω πρόσφατων γεγονότων αποφασίστηκε αυτό, διότι δεν μιλάμε μόνο για τους αρωτές σώματος, μιλάμε για την ασφάλεια της αεροπλοείας ως σύνολο. Οι σαρωτές σώματος είναι ένα από τα θέματα, αλλά είναι ένα ευρύτερο θέμα αεροπλοείας. Ε, δηλαδή, ε, μιλάμε για θέματα ασφαλείας και θα συμπεριλάβουμε και το θέμα της μεταφοράς εμπορευμάτων. Επειδή υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες επιτροπές, ζητήσαμε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Επιτροπή Πολιτικών ε, Ελευθεριών να συμμετάσχουν. Ο κύριος Κίρκοπ εκπροσωπεί την Επιτροπή, όχι Έχω δύο συντονιστές που βρίσκονται πάνω από μένα από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ο κύριος Βος είναι εδώ και νομίζω ότι έχει προτεραιότητα. Θέλω κι εγώ να πω κάτι ως συντονιστής, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί συντονιστές από τη ε, ΛΥΜΠΕ και δεν νομίζω ότι είναι δική μου αρμοδιότητα. Αν θέλετε μπορώ να το κάνω εγώ, αλλά υπάρχουν ε, μερικοί πάνω από εμένα. Εντάξει, συνέχισε, Και εάν ε, οι πολιτικές ελευθερίες, οι δημόσιες ελευθερίες ή το περιβάλλον θέλουν το λόγο, τότε θα λάβω υπόψη την επιχειρηματολογία τους. Θα δω τι θα γίνει με το χρόνο που έχουμε ε, διαθέσιμο. Τίμωθη, θα ήθελα εσύ να αρχίσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο μου είστε αρεστός, αλλά είστε ο πρόεδρος και γνωρίζω τις ε, ότι έχετε τον πρώτο λόγο. Έχετε δίκιο από, πλευρές, από πλευράς ΛΥΜΠΕ. Μιλάμε για ένα ευρύτερο τομέα ασφάλειας, διότι οι σαρωτές σώματος είναι ένα στοιχείο της ασφάλειας και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ μας ενδιαφέρουν τα θέματα ε, ατομικών στοιχείων, εξασφάλισης τους και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε μία εναρμονισμένη προσέγγιση και στις σχέσεις μας με τα άλλα μέρη του κόσμου, διότι μιλάμε για διεθνείς μεταφορές, το θέμα σχετίζεται με τις ΗΠΑ που όπως γνωρίζετε έχει εισαγάγει τις δικές του διευθετήσεις που εμείς ακολουθήσαμε μέχρι ενός σημείου και τώρα γίνεται μία συνάντηση αργότερα μέσα στο μήνα στη Ουάσιγκτον ε, ως με τους ρυθμιστές αεροπλοείας, όπου το θέμα του συντονισμού θα συζητηθεί. Ελπίζω να φτάσουμε σε μία λογική σε ένα λογικό συντονισμό, διότι όπως είπε και ο εισηγητής σας, δεν υπάρχει ομοιομορφία στην προσέγγιση. Βεβαίως η ομοιομορφία είναι πρόβλημα, διότι το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ είπε ότι οι επιβάτες θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτή τη στρωματοποίηση ασφάλειας. Έτσι θα υπάρχει μια δειγματοληπτική διαδικασία, έτσι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν οι επιβάτες. Και αυτό το θεωρεί ισχυρό πλεονέκτημα το Υπουργείο Εσωτερικών. Ξέρετε πώς έχει το θέμα των ε, σαρωτών σώματος. Στο Μάντσεστερ έχουμε προβάλει ε, ένα δελτίο, ένα ερωτηματολόγιο όπου πολλοί προτιμούν τους σαρωτές σώματος από την ψηλάφιση. Και νομίζω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε ένα πολυστρωματικό σύστημα ασφάλειας, αλλά θα πρέπει να ξέρουν οι επιβάτες ε, τι τους περιμένει ή τι να περιμένουν. Πιστεύουμε ότι το θέμα καταπάτησης του ιδιωτικού χώρου των ατομικών δικαιωμάτων, ποιος θα ελέγχει τις εικόνες και τι γίνεται μετά με τις εικόνες αυτών των σαρωτών, ποιος αποκλείεται από αυτό τον έλεγχο, για ποιους λόγους και βεβαίως υπάρχει και το θέμα της υγείας Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη χρήση αυτού του εξοπλισμού. Και τέλος, μας ενδιαφέρει το κόστος. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν κέρδη μετά από πολύ καιρό. Δηλαδή, ποιος φέρει το φόρτο, τα αεροπλάνα, τα κράτη, οι επιβάτες ή οι αεροπορικές εταιρείες. Ποιος θα αναλάβει το κόστος αυτών των μέτρων ασφαλείας διότι θέλουμε να υπάρχει ασφάλεια 100% και είμαστε ρεαλιστές και γνωρίζουμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει 100% αλλά ποιος θα καταβάλει το αντίτιμο και ποια είναι τα όρια σε σχέση με την καταπάτηση ατομικών δικαιωμάτων. Αυτά τα θέματα απασχολούν τη ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστούμε κύριε Κέρκοπ. Μια σύντομη παρατήρηση. Η Επιτροπή αυτή έχει πολύ ισχυρέ απόψει ω προ το ποιο θα επιβαρυνθεί το κόστο. Το θέμα είναι ενισχυμένη ασφάλεια. Άρα, πάρα από αυτή που είναι φυσιολογικά αποδεκτή, θα πρέπει να καταβάλουν το κόστο από τα κράτη-μέλη. Αλλά βέβαια φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη έχουν τελείω διαφορετική άποψη σε σχέση με το θέμα αυτό. Και τώρα πηγαίνουμε στου κοιόδη ηγητέ από την Επιτροπή Μεταφορών. Σα ζητώ να είστε στον πιο σύντομοι, αυτό είναι ο κατάλογος αγορτών μέχρι στιγμή. Θα κάναμε μαθηματικά να δούμε. Πρώτος ο κύριο Φλάκενστάιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, γνωρίζουμε όλοι ότι η απόλυτη ασφάλεια δεν υφίσταται. Υπάρχει λίγη ασφάλεια. Ναι. Αλλά μην δημιουργούμε την εντύπωση ότι η ασφάλεια ε, μπορεί να υπάρξει και να εξασφαλιστεί 100%. Κατά δεύτερον, έχουμε ανάγκη ενός συστήματος ασφάλειας ολοκληρωμένου. Γι' αυτό συμφωνώ με τον εισηγητή που είπε ότι η αποστολή, αυτή η εντολή την οποία έχουμε αναλάβει πρέπει να διευρυνθεί. Γιατί πρέπει πάντα να λαμβάνουμε νέα μέτρα σε ό,τι αφορά τους ε, ταξιδιώτες ε, στα αεροπλάνα, ενώ σε επίπεδο εμπορευμάτων εκεί φαινόμαστε ότι πραγματικά χρονοτριβούμε γιατί στις ε, αέριες, εναέριες μεταφορές ε, θα πρέπει οι ταξιδιώτες να αγδίνονται μέχρι τα σόρουχα, αν επιτρέπετε την έκφραση, ενώ στις δρομικές μεταφορές το καν γίνεται σχετικός λόγος. Τρίτο ερώτημα, αρχικό. Έχουμε ανάγκη ευρωπαϊκών λύσεων. Αυτό έχει αναγνωριστεί από, και από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό ε, Συμβούλιο που προείσταται των συναντήσεων του Συμβουλίου. Είναι απαραίτητο αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά την ε, ε, αποτίμηση του κινδύνου θα πρέπει να ενισχυθεί στην Ευρώπη. Θα πρέπει να υπάρχουν πολύ πιο ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αλλά τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής όταν ετέθη το ζήτημα αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα τους ορωτές, τους ορωτές σώματος καταρχάς γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να απελευθερωθούν της υποχρέωσης να χρήσεις των ε, σαρωτών. Εάν υποχρεωθούν θα πρέπει να έχουμε ισότιμες συνθήκες και μεταξύ αυτών βεβαίω την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που δεν θα πρέπει να μεταδίδονται, ε, που δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται, και που δεν είναι θα πρέπει να υπάρχουν συνέπειες αρνητικές σε ό,τι αφορά την, απο... την υγεία των ταξιδιωτών και θα πρέπει το σύστημα αυτό να είναι πάρα πολύ γρήγορο ώστε να αντικατασταθούν τα εφιστάμενα συστήματα. Για να υπάρχει ένας λογικός κανονισμός χρηματοδότησης ό,τι αφορά τους ερωτές αυτούς, θα πρέπει το Συμβούλιο να συμφωνήσει πάνω σε ένα σχέδιο οδηγία για την ε, ασφάλεια των αέριων μεταφορών και του κόστους που θα πρέπει να επιμεριστεί. Βεβαίως, οι επιβάτες θα πρέπει να καταβάλουν τα σχετικά έξοδα σε ό,τι αφορά την ίδια ασφάλεια. Αλλά όταν μιλάμε για ε, μεταφορά, αέρια μεταφορά φορτίων, δεν υπάρχει πλέον ε, επιβάτης. Άρα όλα τα θεσμικά όργανα, τα υπουργεία, τα Εθνικά Υπουργεία, η Επιτροπή μας είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια λογική σχέση κόστους που θα επιμεριστεί. Και είμαι πεπισμένος ότι το ίδιο θα ισχύσει και για τους προσωπικούς ερωτές σώματος. Ένα τελευταίο σημείο. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια αξιολόγηση και ας δούμε πλέον τότε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Προς το παρόν υπάρχουν αυτοί οι προσωπικοί σαρωτές σώματος στο Άμστερνταμ, το Παρίσι και το Μάντσεστερ. Ο καθένας προσπαθεί να κάνει και να λειτουργήσει κάτω δοκού, γιατί για παράδειγμα στο Μιλάνο καταργήθηκαν, στο Αμβούργο ξαναξεκίνησαν, πλέον είναι καιρός να θέσουμε κοινού στόχους και να δράσουμε κατά τον ίδιο τρόπο, ώστε όλοι να έχουμε πραγματικά αναλογική προσέγγιση. Υπό αυτή την έννοια, όντως μπορούμε να φανταστούμε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να εισάγουν τα, τους προσωπικούς αρωτές, αλλά δεν μπορούμε αυτό να το καταστήσουμε υποχρέωση. Ναι, δεν έχω δει το σχετικό ε, χρόνο. Πέντε λεπτά θα είναι για τα σκιώδεις ε, ε, εισηγητές και τρία για τα μέλη της Τέσσερα λεπτά για την ομάδα των Πρασίνων. Κυρία Μάιστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για όλη την προπαρασκευαστική εργασία που έκανε και την ε, συζητήση που είχαμε ήδη. Πρόκειται εδώ για την ασφάλεια στι ενέργειε μεταφορέ και όπω πολύ στα ελέγχθη δεν υπάρχει ασφάλεια 100%. Ταυτόχρονα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το οποίο διαθέτουμε αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ χαμηλό σε ό,τι αφορά θέματα ασφάλεια. Υπάρχει τεχνολογία που θα μα επέτρεπε να διασφαλίσουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Βέβαια, ο τομέα αέριων μεταφορών φορτίων, εμπορευματικών μεταφορών, όντω είναι κάτι το οποίο διακυβεύεται. Ήρθαν πάρα πολλοί συμβασμοί τελευταία και βλέπουμε ότι το πακέτο από το, με τα μεταφορική UPS που εστάλει στη Μέρκελ είδαμε ότι ήταν, είχε εκρηκτικά και δεν είχε ανακαλυφθεί. Άρα είναι μια απόδειξη του ότι πάρα πολλά όργανα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και εξοπλισμοί δεν είναι καθόλου ε, αποτελεσματικοί. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις εμπορευματικές μεταφορές, ε, όπω μεταφορές, όπως ήδη ελέγχεται τον προηγούμενο μιλητή, ε, υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός πακέτων. Όταν υπήρχε το, σκό, το νέφος της ε, ε, σκόνης, πάλι υπήρχαν πάρα πολλά ζητήματα και πάρα πολλά, αν θέλετε, πολύτιμα τα οποία είχαν σταλεί και τα οποία δεν ήταν. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν, να δούμε ποια μέτρα, τα μέτρα τα οποία θα εισαχθούν, να μην καθυστερούν σε όλες τις διαδικασίες για τα αεροδρόμια, τώρα που μιλάμε εδώ, πολύ συχνά έχουμε μιλήσει κατά κύριο λόγο για σαρωτέ που επουδενή δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια. Το ίδιο πρέπει να θέσουμε το ερώτημα σε ποιο μέτρο έχουμε ανάγκη περισσότερο προσωπικού. Ε, το αεροδρόμιο Τελαβέβ, για παράδειγμα, είναι το πλέον ασφαλέ στον κόσμο, αλλά εκεί υπάρχει ευθύ εξ αρχή μια αρνητική διάκριση που λέει ότι όσοι είναι Άραβε ηλικία 20 έως 50 είναι εξορισμού ε, Άρα πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό, αν θέλετε, έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε όλο το απαραίτητο ε, προσωπικό και πόσοι θα υπόκεινται σε σχετικό έλεγχο. Οι σαρωτές λοιπόν, όντως τα στοιχεία ε, παίζουν ένα ρόλο, τα πικτογράμματα είναι σημαντικά, τα, ε, επίσης δεν θα πρέπει να διακυβεύεται η υγεία των αξιδιωτών που παίρνουν τους σαρωτές αυτούς και επίσης πρέπει να ξέρουμε περί ποιες τεχνολογίε μιλάμε. Ακτίνες χ, κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το δεχτούμε εμείς οι ακτίνες Χ μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για ιατρικούς σκοπούς και πάλι τίφτε ζήτημα. Υπάρχουν άλλα όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται, τα οποία όμως ακόμα δεν είναι απολυτελεγμένα. Τι γίνεται με τους ε, σαρωτές, ε, ε, τι ασφάλεια έχουμε με τους σαρωτές, πολύ περισσότεροι από τώρα ίσως. Πρέπει όμως να δούμε οπωσδήποτε τους κινδύνους υγείας που ενδεχομένως υπησέρχονται. Θα πρέπει να ελέγξουμε πώς ε, θα, ποια θα είναι και η ταχύτητα λειτουργίας, πόσα άτομα θα παίρνουν από τους ορωτές ε, ανά ώρα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια. Στη συνέχεια βέβαια το θέμα του κόστος. Ποιο θα, θα, θα πληρώσει για όλα αυτά. Μπορούμε να το εφαρμόσουμε για τις χειραποσκευές, τους αρωτές αυτούς. Όπως θα το επιθυμούσαμε ίσως. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, όλους τους παράγοντες, να τους αξιολογήσουμε και να λάβουμε σχετική απόφαση. Τι γίνεται με την ενδεχόμενη χρήση εκρηκτικών. υπάρχουν σχετικές εμπειρίες από άλλα δρόμια. τι επιτρέπεται πριν από τους διάφορους ορωτές. Δεν υπάρχει να υπάρχει ενιαία λύση σε όλα αυτά, αλλά πρέπει να υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση, μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΕ. Και έχω συγκεκριμένα ερώτημα να απευθύνω στην Επιτροπή σχετικά. Πέρσι έγινε συζήτηση περί υγρών και της ε, χρήσης και μεταφοράς ε, των προϊόντων από duty free από τους σαρωτές. Νομίζω ότι το πλέον τα υγρά προϊόντα μπορούν να περάσουν από τους σαρωτές. Δεν ήταν απόφαση αυτό του, αυτή του Κοινοβουλίου, αλλά ήταν, αν θέλετε, μια μετάφραση αυτού που θέλαμε να επιτύχουμε, δηλαδή να εξασφαλίσουμε μια ενιαία συσκευασία. Η ερώτημα λοιπόν είναι ποια είναι η τεχνολογική θέση τώρα, ποια είναι η τελευταία τεχνολογία που υπάρχει ό,τι αφορά του ορωτέ. Τώρα επιτρέπεται η μεταφορά ε, υγρών στην καμπίνα. Την Μπέργκερ και του πράσινου. Ευχαριστώ πολύ για την εναρμόνιση αυτών που πρέπει να χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη συμφωνώ απολύτως. Ε, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι θα υπάρχει δυνατότητα να δεχθεί κανείς τη χρήση των σαρωτών ή όχι. Τα αποτελέσματα που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή για τους σαρωτές σώματος δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά όσο θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε η βιομηχανία κρατάει, ε, ο, ο, χρόνος, ο χρόνος παρατείνεται και σε πάρα πολλές περιπτώσεις γίνεται, και, ακολουθείται και η διαδικασία της ψηλάφισης και γίνονται και πολλά λάθη κατά την ανείχνευση και όλη η διαδικασία απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Αν δεν έχουμε, ε, πρέπει να αναπτύξουμε τις υποδομές, να τις διπλασιάσουμε, να τις τριπλασιάσουμε, διότι αν χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα για τον έλεγχο κάθε επιβάτη, οι καθυστερήσεις θα είναι τεράστιες. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις θα υπάρξει πρόβλημα. Το συζητήσαμε στην Επιτροπή Μεταφορών το θέμα αυτό κατ' επανάληψη. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε να ρυθμιστεί το όλο θέμα από οικονομική άποψη. Και έρχομαι τώρα σε ένα άλλο σημαντικό σημείο. Αν πούμε ότι η χρηματοδότηση δεν έχει ακόμα ρυθμιστεί, ότι τα στοιχεία που λαμβάνουμε δείχνουν ότι έχουν γίνει λάθη κατά τη χρήση, λάθη ανείχνευσης, ίσως χρειαστεί να προβλέψουμε κάτι άλλο. Υπάρχει μια πραγματικότητα όμως την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη. Οι άνθρωποι σήμερα δεν δέχονται, δεν θέλουν να αποδεχθούν τα τεχνικά σύνορα. Δεν μπορεί να ανοιχνευθούν από τους αρετές όλα τα χημικά προϊόντα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να την αποδεχθούμε και να την έχουμε υπόψη μας να ξανασκεφτούμε σοβαρά το θέμα και να δούμε πώς τίθεται αυτό σε σχέση με την ε, απόφαση ενδεχομένω να ζητήσουμε μία παρέκκληση. Μπορεί ένα κράτος ε, να αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσει αυτά τα συστήματα, ναι ή όχι, για τα εμπορεύματα, για τα φορτία. δεν μιλάμε μόνο για τη μεταφορά πολύτιμων αντικειμένων. Όταν προέκυψε η κρίση λόγω της ε, ηφαιστιακής στέφρας, είδαμε μεταφορά οποροκυπευτικών από την ε, Αφρική. Και θέλω να διατυπώσω και άλλη μια ερώτηση. Αυτή την εποχή Ίσως πιστέψετε ότι μιλάω υπέρ του δικού μου πανεπιστημίου, αλλά αυτή την εποχή ε, ε χρηματο... Ε, ε, αναπτύσσεται ένας αεριοχρωματογράφος που επιτρέπει την ανείχνευση χημικών συνδυασμών και ενώσεων με βάση την οσμή τους. Μήπως λοιπόν αυτή είναι μια τεχνολογία που θα έπρεπε να την εξετάσουμε με μεγαλύτερη προσοχή, διότι μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη, χρήσιμη για, τους, για επιβάτες και για τα εμπορεύματα. Διότι αν δεν κάνουμε κάτι για, το, για τα εμπορεύματα, δεν βλέπω για ποιο λόγο. Θα προσθέτουμε ε, ελέγχους για τους επιβάτες αγνώντας τα εμπορεύματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια γρήγορη απάντηση στην κυρία Μάισνερ πρώτα. Το γεγονό ότι δεν μπόρεσα να έρθω σε επαφή με τον εισηγητή οφείλεται σε, μια, σε ένα ταξίδι μελέτη που έκανα ε, στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ. Ελέγχθηκα, με, ελέγχθη, με ελέγξαν από την κορφή μέχρι τα νύχια. Αυτό πρέπει να σας πω για το περιεχόμενο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό ο εισηγητής να επιστήσει την προσοχή στη... σε αυτά τα οποία ισχύουν στη Δύση θα χρειαστεί να διαθέσουμε χρήματα και προσωπικό και το κάνουμε αυτό διότι αντιμετωπίζουμε την απειλή της τρομοκρατίας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Να πούμε δηλαδή και να τονίσουμε ότι αντιμετωπίζουμε, αντιμετωπίζουμε τρομοκρατικές απειλές με, από οργανώσεις όπως η Αλκάιντα. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Και πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη το γεγονός ότι δεν έχουμε ασφάλεια 100%. Αυτό είναι αδύνατο. Η ασφάλεια είναι κάτι παραπάνω από έναν σαρωτή σώματος. Λέμε, λένε πολλοί, ε, χρησιμοποιήσουμε σαρωτή σώματος και το πρόβλημα θα έχει λυθεί. Μα δεν είναι έτσι. Αυτό που χρειάζεται είναι ανταλλαγή πληροφοριών, ανταλλαγή στοιχείων, συνεργασία ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές για να περιορίσουμε, να περιορίσουμε την απειλή ο σαρωτή σώματος είναι ένα μόνο στοιχείο όλης αυτής της διαδικασίας. Το σαρωτή σώματος πρέπει να τον προσθέσουμε στο οπλοστάσιο που διαθέτουμε για την καταπολέμηση τρομοκρατίας. Θα είναι αυτό ένα μέσο ανάμεσα σε άλλα ο σαρωτή σώματος. Δεν πρέπει όμως να είναι η χρήση του υποχρεωτική. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα για τον επιβάτη να αποφασίσει αν θα περάσει από το σαρωτή σώματος ή θα ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία για τον έλεγχο. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Και τα θέματα υγείας. Πολύ σωστά είπατε ότι πρέπει να περιορίσουμε τη χρήση των ακτίνων Χ. Δεν νομίζω ότι στη σήμερα ημέρα υπάρχουν αεροδρόμια που χρησιμοποιούν ακτίνες Χ για τους ελέγχους. Αν ναι, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το αντιμετωπίσουμε. Και πρέπει να μην ακούμε αυτά τα παραμύθια για, τους, για τους, τα μηχανήματα της δεύτερης γενιάς που επιτρέπουν, επιτρέπουν ε, να βλέπει κανείς μια πολύ ολοκληρωμένη εικόνα του ατόμου με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η ατομική του ελευθερία. απλώς ε, αυτός ο σαρωτής, οι σαρωτές δείχνουν μία επιτρέπουν ενδεχομένω να εντοπιστεί κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να, είναι, να βρίσκεται εκεί, χωρίς όμως να δίνουν μια σαφή εικόνα του, του σώματος του ατόμου που υφίσταται τον έλεγχο. Στο παράρτημα που θα ετοιμάσουμε θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τις ε, μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτά ήθελα να σας πω. Θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε, αλλά πιστεύω ότι αυτά τα σημεία που έθιξα είναι σημεία κλειδί. Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε που τηρήσατε το χρόνο σας. Ο κ. για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. οι αεροπορικές εταιρείες θέλουν συνεχώς να περιστέλουν το κόστος, άρα είναι ένα καλό βήμα να ενισχύσουμε την ασφάλεια. Η εναρμόνιση είναι σημαντική βεβαίως, αλλά ποιο το πρόσθετο τίμημα και πρέπει βέβαια να μιλήσουμε περί των εμπορευματικών μεταφορών επίσης. Η ασφάλεια και η ε, εξασφάλιση του απόρριτου των προσωπικών στοιχείων είναι δύο αντιφατικές έννοιες. Και υπάρχουν και θέματα υγείας, συν παρακράτηση προσωπικών στοιχείων προσπαθώ να χαμογελώ όταν παίρνω από έλεγχο, γιατί δεν ξέρω τελικά τι περνάω και τι αποθήκευση στοιχείων θα υπάρξει. Και προσλέπω αν θέλετε, βλέπω αυτές τις ε, φωτογραφικές εικόνες, οι οποίες κάπου αποθηκεύονται, που ίσως καταλήξουν κάποια στιγμή και σε κίτρινο τύπο. Πολύ, ε, πολύ γοητευτικά θα είναι τα, τα πρωτοσέλιδα που θα δούμε. Τι, τι εξετάζουμε αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω ακριβώς. Τι αναζητούμε, μεταλλικά στοιχεία, υγρά, πλαστικά, τι αναζητούμε από τους ελέγχους αυτούς. Χημικές ουσίες, όπως ανέφεραν συνάδελφοι. Είναι αλήθεια ότι λίγα μόρια μπορούν να ανοιχνευθούν μόλις απειροελάχιστα με χρωματογράφο. Εάν θέλετε μπορούμε να επισέλθουμε και σε λεπτομέρειες. Τεχνικές λύσεις. Έχουμε ε, για τα διάφορα μέταλλα διάφορους ε, ανιχνευτές ε, μέσω ακτινοβολίας. Τα έχουμε όλα αυτά. Όμως, ποιο θα είναι το πρότυπο, ποια θα είναι τα πρότυπα που θα εφαρμοστούν εδώ. Θα είναι η ασφάλεια δεδομένων. Τι άλλο. Δεν γνωρίζω ακριβώς και ως συνήθως επανερχόμαστε στα 120 ml που είναι ένα αυθαίρετο κατόφλι που έχει τεθεί οροφή, αν θέλετε, για τα υγρά. Κάποια αεροδρόμια σα αναγκάζουν να βγάζουν τα παπούτσια, αλλά όχι. Κάποιε φορέ πρέπει να περάσουμε μέσα από ακτίνε χ, σε άλλα όχι. Δεν υπάρχει τρόπο να εξασφαλίσουμε και να ενισχύσουμε την ασφάλεια κατά αυτόν τον τρόπο. Σα διαβεβαιώ. Ευχαριστώ. Και τώρα πάω το επόμενο ανατρίλεπτο. Ξεκινάμε με τον κύριο Γκρό. Έχω ένα κατάλογο 14 αγοριτών. Λοιπόν, τρία λεπτά ο καθένας. Και θα είμαι πάρα πολύ αυστηρό στου ε, φίλου από, από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών που δεν με ξέρουν πραγματικά. Μπορώ να είμαι πάρα πολύ σκληρό με το σφυράκι αυτό. Κύριε Γκρό, τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βλέπω το πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την εξέλιξη τεχνολογίας την ε, ε, εφαρμοσιμότητα, την αξιοπιστία και την αναγνώριση της εκλογίας. Θα, προ, θα εδώ και την εναρμόνιση και θα έλεγα ότι θα έπρεπε να να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια βασικά κριτήρια σε ό,τι αφορά την αναγνώριση. ώστε να έχουμε πραγματικά αξιόπιστα στοιχεία ανεξαρτήτως πηγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει κάτι να κάνει και να λάβει δράση. Κατά δεύτερον, εδώ πρόκειται για τη διαφορά μεταξύ των υποχρεωτικών μέτρων και τη ελευθερία κάθε κράτου μέλου να λάβει τα δικά του μέτρα. Και καταλήγουμε αυτό σε ό,τι αφορά θέματα χρηματοδότηση, που είναι πάρα πολύ μακρά η όλη συζήτηση. Είμαι της άποψης και νομίζω είναι κοινοβουλευτική άψη ότι σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση υποχρεωτικών μέτρων θα πρέπει να οι εθνικές αρχές να έχουν εξουσία και να λάβουν δράση. Όμως θα πρέπει να έχουμε μέτρα τα οποία θα εφαρμόζουν τις βασικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τα θέματα ελευθερία, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα μέτρα υγείας. Πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση στην προσέγγιση και για αυτό το λόγο από κοινού μπορούμε να, κάνουμε προ... να σημειώσουμε πρόοδο. Τέλος, δεν πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο χρειάζεται να εμπλακεί στις μικρές λεπτομέρειες κάθε τεχνολογικής ε, ε λεπτομέρειας αυτών των θεμάτων. Πρέπει να διασφαλίσουμε τις βασικές ελευθερίες που δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται από την υιοθέτηση τη σύγχρονη τεχνολογία. Και εξακολουθεί να εκκρεμεί ένα ερώτημα. Είναι το Συμβούλιο πρόθυμο και έτοιμο να αναλάβει συντονισμένη προσέγγιση σε αυτό, ναι ή όχι. Αν δείτε τα πόσα σημαντικά θέματα διακυβεύονται σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, θα έλεγα ότι θα έπρεπε ευθύ εξ αρχή να θέσουμε το ερώτημα. Το Συμβούλιο, τα 27 κράτη-μέλη είναι πρόθυμα να ακολουθήσουν αυτή την πορεία. Αξίζει να καταβάλουμε όλες αυτές τις μεγάλες προσπάθειες. Ή το Συμβούλιο απλώς θα κάνει το κεφαλιού του. Εγώ θέλω να ζητήσω ενίσχυση του Ευρωπαϊκού, Κοινού Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και βέβαια δεν θα προωθήσουμε τη θέση μας λειτουργώντας ξεχωριστά από τη ΣΥΠΑ. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Άλκεντο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Σίγητη για την εισαγωγή του και για την ετοιμότητά του και την προσπάθεια επίτευξης κάποιας συνένεσης. Σίγουρα στην έκθεση αυτή θα πρέπει να εστιάσουμε πάνω στην έκθεση της Επιτροπής για τους αρωτές, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να δούμε τα θέματα ασφάλειας των εναέριων μεταφορών, τόσο επιβατών όσο και εμπορευμάτων και να έχουμε συνολική προσέγγιση. Δυστυχώς ε, δεν έχουμε προληπτική δράση, μονίμως αντιδρούμε εκ των υστέρων σε ένα συμβάνι, σε μια απειλή και τότε θέλουμε και είμαστε έτοιμοι να εισάγουμε νέα μέτρα. Προσθέτουμε λοιπόν μέτρα επί των μέτρων και τελικά όλος ο μηχανισμός είναι εξαιρετικά δαπανηρός και βαρύς. Το θέμα είναι να εξορρομπήσουμε μια προληπτική δράση ασφάλειας και θα πρέπει να υπάρξουν κατάλληλοι πόροι που θα επιτρέπουν ευελιξία και διαβούλευση. Πρέπει να εστιάσουμε και στα θέματα ε, αποτελεσματική χρηστή διακυβέρνηση, αλλά και εξασφάλιση προσωπικών στοιχείων. Θα πρέπει να δούμε τους μακροπρόθεσμου στόχου τις τεχνολογικές εξελίξεις, την ασφάλεια, την βιομηχανική πολιτική που θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη και βέβαια όσο αυτό είναι δυνατόν θα πρέπει να έχουμε μια ενιαία προσέγγιση, μια ενιαία πολιτική. Θα πρέπει να αποφύγουμε την λήψη μονομερών μέτρων από τα κράτη-μέλη. Αυτό θα πρέπει πάση θυσία να το αποθαρρύνουμε. Αλλά ταυτόχρονα, όπως ε, ήδη ελέγχθη, θα πρέπει να σκεφτούμε και τη σχέση μας με τις ΗΠΑ. Υπάρχει μια σχετική συμφωνία για την αεροπλοεία και θα συσταθεί και μια κοινή επιτροπή όπου θα συζητούνται όλα αυτά τα ζητήματα. Σε αυ περί αυτών των διάσημων σαρωτών σώματος συμφωνώ με αυτό που είπαν πάρα πολλοί ομιλητέ. Χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για νομικούς λόγους. ένα κράτος μέλος μπορεί προσωρινά πάντα να χρησιμοποιήσει τα μέτρα αυτά ή να χρησιμοποιήσει άλλα, αλλά χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τα θέματα δημόσιας υγείας, προστασία προσωπικών δεδομένων, κόστους αλλά επίσης και τα θέματα κατάρτισης. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους που θα ε, χειρίζονται τους αρωτές αυτούς. Εστιάζουμε πάρα πολύ πάνω στα μηχανήματα, αλλά τι γίνεται με, αυτούς, με τους χειριστές των μηχανημάτων. Πρέπει να το σκεφτούμε. Και επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι μια, η αποτελεσματική τεχνολογία εξελίσσεται. Οι σαρωτές λοιπόν σώματος μπορούν επίσης και εξελίσσονται. Διαφωνώ με την άποψη του κ. Βαντέλεν που λέει ότι στο προσάρτημα ότι πρέπει να είμαστε δυνατόν πιο ανοιχτοί. Πιστεύω ότι αν προκύψει κάτι καινούριο θα πρέπει να το αξιολογούμε πρώτα. Θα πρέπει να δούμε και σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση προσωπικών στοιχείων. Προσβλέπω λοιπόν σε καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μπιλμπάου τρία λεπτά. Μπιλμπάου είπε. Θα ήθελα να σας πω ότι συμφωνώ ότι οι σαρωτές είναι ένα στοιχείο επιπροσθέτως στο σύστημα ασφάλειας, αλλά η τρομοκρατία προτρέχει, βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά από εμάς. Γι' αυτό θα πρέπει να προτρέχουμε και εμείς δηλαδή όχι να βρίσκουμε εμβαλωματικές λύσεις. Θα πρέπει να εξισορροπήσουμε την κατάσταση μεταξύ ασφάλειας, υγείας και υγείας, ιδιαίτερα των χειριστών των σαρωτών. Και θα πρέπει να είμαστε σαφείς για το πώς θα διαχειριστούμε τα δεδομένα τη στιγμή που θα τεθούν σε εφαρμογή οι σαρωτές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί συμφωνώ με την διαχείριση δεδομένων, γιατί μίλησε για ε, το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να δούμε τι θα γίνει και με τις εγγραφές στους αρωτές και με τους χρωματογράφους. Νομίζω ότι βρισκόμαστε κάπως πίσω, διότι υπάρχουν που θέτουν σε εφαρμογή ήδη τα συστήματα που θεωρούν πιο αποτελεσματικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να προβάλλουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το θέμα των σκάνερ και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την καινοτομία και την τεχνολογία έτσι ώστε να έχουμε μια αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών μελών μέσω των τεχνολογικών κέντρων και πανεπιστημίων για να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα συστήματα και να προτείνουμε, να προβάλλουμε μία ευρωπαϊκή πρόταση που θα μας διευκόλυνε στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και τις άλλες χώρες και θα μπορούσαν να έχουν εμπιστοσύνη σε μας και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Χάνουμε πολύ χρόνο, θα πρέπει να συντονιστούμε με τα τεχνολογικά κέντρα και να φτάσουμε σε ένα ευρωπαϊκό ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Μιλάμε για τις δαπάνες, για το συνολικό κόστος. Ε, μας ρωτάτε πόσο θα στοιχήσει, μα πόσο μας στοιχίζει και η παρούσα ασφάλεια Ας πάρουμε το αεροδρόμιο των ε, Βρυξελών. Η ασφάλεια στοιχίζει τόσο, ένα σαρωτής στοιχίζει τόσο. Άρα θα δούμε ποια είναι η διαφορά. Θα πρέπει να εργαστούμε με στόχους που θα μας οδηγήσουν σε μια μεγαλύτερη σαφήνεια. Είμαι υπέρ της ε, ευρωπαϊκής προσέγγισης και είμαι και υπέρ των σαρωτών. Διότι με έχει κουράσει πια η επιθετικότητα των ε, χειριστών των μηχανημάτων που πρέπει να με ψηλαφίσουν κάθε φορά στο αεροδρόμιο. Πραγματικά με έχει κουράσει αυτό το σύστημα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αύριο ταξιδεύοντας στο Σκύπολ θα μπορούσατε να υποβάλλετε συγκεκριμένες ερωτήσεις και προς τις αρχές η επόμενη ομιλήτρια. Είχαμε μία πολύ χρήσιμη συζήτηση, δεν χρειάζεται να πω τα ίδια. Πολλοί εξέφρασαν ανησυχίες, διότι μιλάμε για ένα επιπρόσθετο στοιχείο, το οποίο δεν είναι πανάκια. Μπορούμε να έχουμε σαρωτές παντού. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτός ο εξοπλισμός θα σταματήσει έναν τρομοκράτη. Νομίζω όμως ότι ζούμε σε έναν πραγματικό κόσμο όπου οι σαρωτές είναι υποχρεωτικοί και στο Σκύπολ και στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε μερικά άλλα αεροδρόμια. Από τη δική μου πλευρά πιστεύω ότι υπάρχει το θέμα της τεχνολογίας αλλά και το θέμα της υγείας σε σχέση με τις ακτινοβολίες, με τις ακτίνες Χ. Υπάρχει ε, το χιλιομετρικό κύμα, το οποίο ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, διότι ο εξοπλισμός αυτός δεν θα πρέπει να έχει αρνητικές επιπτώσεις. Δεν μιλάμε μόνο για τους επιβάτες. Υπάρχει προσωπικό που χειρίζεται αυτά τα μηχανήματα καθημερινά. Εμείς ταξιδεύουμε δύο φορές τη βδομάδα. Θα πρέπει λοιπόν ο εξοπλισμός αυτός να μην έχει επιπτώσει στην υγεία. Το θέμα εφήγει και ως προς τις εικόνες, τους χρωματογράφους. Νομίζω θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την καλύτερη δυνατή τεχνολογία. Μιλάμε για τα υγρά, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε και Στη συνέχεια έχουμε κάποιον από την Ιεμένη, ο οποίος μεταφέρει ό,τι θέλει μέσω φορτίων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν σαρωτές και για τα φορτία, όχι μόνο για τους επιβάτες, αλλά αυτό ε, αφορά μια γενικότερη επαγρύπνηση. Θα πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστές για το που βρισκόμαστε. θα πρέπει να βρούμε μία εξισορροπημένη λύση. Διότι βρέθηκα στην άλλη πλευρά του ζητήματος, ε, είχα καταρτιστεί για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και όταν μιλάτε στο προσωπικό του αεροδρομίου, έχουν μία εξισορροπημένη προσέγγιση, ξέρουν πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν και να προσεγγίσουν το ζήτημα. Αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε κι εμείς. Θα υποστηρίξουμε τον εισηγητή μας και τους σκιώδεις και ελπίζω να έχουμε μία πολύ εξισορροπημένη προσέγγιση. Τέλος, μετά την 10η Σεπτεμβρίου ε, μιλούσαμε για τις χώρες ΙΚΑΠ και δεν τον εφάρμοσαν τον κανονισμό μόνο οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι περάσει εδώ θα έπρεπε να βοηθήσει και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες έτσι ώστε να έχουμε ομοιόμορφη προσέγγιση. Next is uh, Mr. Diaz from Civil Liberties. Ο κύριος... Ο Δίας από τη ΛΥΜΠΕ. Σας ευχαριστώ. Ε, συμμετέχω στην ε, ΛΥΜΠΕ και θα παρακολουθήσω με μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το εγχείρημα. Θα ήθελα να πω ότι ασφάλεια στην αεροπλοεία είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, αλλά ένα αναγκαίο κακό. Ε, η, ως προς τα φορτία, εδώ δεν μιλάμε για πρόσκρουση σε ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε σαρωτές φορτίων, γιατί μπορούν να ανοιχνεύσουν μεταλλικά ε, στοιχεία εκρηκτικά και ούτω καθεξής. Και επίσης το φορτίο σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ανοιχτευτεί το περιεχόμενό του, αλλά χωρίς να υπάρχει θέμα του ότι θίγουμε κάτι ή κάποιον. Μέσα στα πλαίσια της υγείας και της, ε, της υγείας και της ε, ανείχνευσης φορτίων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ορισμένα στοιχεία ίσως μας ενοχλήσουν. Εν πάση περιπτώσει, μας ενδιαφέρει η ασφάλεια και η, ε, η απαλυφή των εικόνων θα πρέπει να είναι άμεση, να καταστρέφονται δηλαδή οι εικόνες αμέσως μετά από τον έλεγχο, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των ατομικών δικαιωμάτων. Οι άνθρωποι με ειδικέ ανάγκες, οι έγκυες γυναίκες, τα μικρά παιδιά θα πρέπει να περνάνε από άλλα ε, μέτρα, τα οποία να μην θέτουν σε κίνδυνο την υγεία. Γιατί πιστεύω ότι η ασφάλεια στο, στον αέριο χώρο είναι πολύ πιο σημαντική γιατί είναι θανατηφόρα εάν φυγούν ή εάν υπάρξουν ορισμένα ε, δύσκολα και στοιχεία τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε ε, θανατηφόρες συνέπειες. Το κόστος είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα διαχρονικά ωφέλη. Αυτό το βλέπουμε και στο Hall» και στο Ισραήλ. Διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ότι τελικά πρόκειται για ένα φτηνό σύστημα και οπωσδήποτε η νομική πλαισίωση θα πρέπει να γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ο κ. Καντάου ήταν εκείνο που είπε ότι έχουμε την τάση να αντιδράμε αρκετά βία για το θέμα αυτό. Στη δεκαετία του 70 στην Ολλανδία υπήρχε μια τρομοκρατική ομάδα η οποία στη διάρκεια ενός έτους ε, κράτησε σε ομοιρία μια ολόκληρη τάξη παιδιών σε ένα τρένο και σκότωσαν 7 άτομα σε μια πρεσβεία. Και δεν θυμάμαι όμως εκείνη την εποχή να εξοπλίσαμε όλες τους παιδικούς σταθμού και όλα τα νηπιαγωγεία με σαρωτέ σώματο. Έχουν λεχθεί πολλά για τις τεχνικές λεπτομέρειες του εξοπλισμού για τον οποίο μιλάμε. Αλλά ίσως πρέπει να δούμε και τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Τι κινεί όλη αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει αυτή τη στιγμή για την κατάργηση των θεωρήσεων, το πρόγραμμα κατάργηση των θεωρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών σε, στα πλαίσια διμερών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και επιμέρους κρατών και υπάρχουν και συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουν, οι ΗΠΑ έχουν έναν κατάλογο ε, προϋποθέσεων ε, ε, έλεγχη ασφαλείας όρια ασφαλείας που πρέπει να επιβληθούν σε όλα τα αεροδρόμια. Αλλά δεν γνωρίζουμε τίποτα για όλα αυτά. Και ίσως αυτά που συζητούμε σήμερα να έχουν ήδη πώς αποφασιστεί και απλά χάνουμε το χρόνο μας. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η ασφάλεια είναι κάτι το σημαντικό για όλους μας. Είναι στα, στα γονίδια μας αυτή η ανάγκη για ασφάλεια. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό το σημαντικό πράγμα και να διαβάσετε μια, ένα κείμενο για τη χρηματοδότηση, για έρευνα στον τομέα της ασφάλειας το, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάρα πολλά χρήματα δαπανώνται για αυτό το σκοπό, για την ανάπτυξη διαφόρων τεχνολογικών λύσεων και χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια. Πρέπει να δούμε ποια συμφέροντα διακυβεύονται εδώ. Εμείς έχουμε συμφέρον και επιθυμούμε να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, αλλά υπάρχουν και τα συμφέροντα της βιομηχανίας, τα οποία δεν είναι απόλυτα διαφανή και τα οποία πρέπει να προσδιορίσουμε πρέπει να στηριζόμαστε σε συγκεκριμένα γεγονότα, όχι σε εικασίες. Το δέμα το οποίο ε, εντοπίστηκε ε, ε, πρόκειται νομίζω για έναν εκτυπωτή ε, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει καθημερινά. Καθημερινά δεν πιστεύουμε στις συνωμοσίε, αλλά είμαστε ε, πολιτικοί και ξέρουμε ότι το, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών απαιτεί 100% σάρωση, ε, και φαίνεται ότι είναι πλέον έτοιμοι να πάρουν αυτή την απόφαση. Αυτό λοιπόν που προέχει να έχουμε πλήρη ενημέρωση για τα γεγονότα και για τα στοιχεία που υπάρχουν. Ο κύριος Ζασάντ. Bardzo Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν είμαι ιδιαίτερα ενθουσιώδης για τους αρωτές σώματος και μπορώ να διαβεβαιώσω εκείνους που έχουν, γιατί συμφωνώ με εκείνους οι οποίοι λένε ότι παραβιάζεται ε, ε, και δεν ξέρω, ε, δεν συμφωνώ με εκείνους που λένε ότι παραβιάζεται η ιδιωτική μας ζωή, διότι και ότι δεν, δεν, δείχνουν, δεν όλα τα χαρακτηριστικά του σώματος, μπορούν να δείξουν ότι κάτι μεταφέρει στο σώμα του ο επιβάτης, αλλά δεν φαίνεται αν είναι πακέτο, ένα t-shirt ή μια βόμβα. Δεν είναι δυνατόν να το διευκρινίσει κανείς αυτό. Και αν κάτι είναι κρυμμένο μέσα στο σώμα, στο, στο στόμα σας παραδείγματο χάρη, ή όταν ε, ε, κρύβονται, τα, όπως την άλλη περίπτωση που είχαν κρύψει βόμβες στο σώμα ενός σκύλου, αυτά δεν εντοπίζονται από το σαρωτή. Ένα σαρωτής ε, κοστίζει πολλά λεφτά χρειαζόμαστε τουλάχιστον καμιά δωδεκαριά σκάνερ σε κάθε αεροδρόμιο. Μιλάμε λοιπόν για μερικά εκατομμύρια ευρώ συνολικά και σε πάρα πολλά αεροδρόμια που είναι πολύ μεγάλα και έχουν πάρα πολλούς αρωτές, τα ποσά φτάνουν στα δισεκατομμύρια. Αν θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι κάτι κάνουμε για το θέμα της ασφάλειας στο Κοινοβούλιο, τότε είναι καλό άλοθη οι σαρωτές. Αλλά δεν θα μας δώσουν την ασφάλεια που χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ κύριε Σασάντ και ευχαριστώ γιατί υπήρξατε σύντομα Κύριε Δανέλη. Πρόεδρε, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι από την εμφάνιση των φαινομένων τρομοκρατίας άρχισε να τίθεται με ένταση ε, το ερώτημα των ορίων μεταξύ της ασφάλειας και της περιστολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και των προσωπικών ελευθεριών. Και βέβαια μαζί άρχισε και ένα κυνηγητό που μας βρίσκει πάντα πίσω από την ευρηματικότητα των επίδοξων τρομοκρατών και από την πρόοδο της τεχνολογίας. Το ποια είναι αυτά τα όρια μεταξύ της ε, διασφάλισης της προστασίας ε, αλλά και της ε, επίσης διασφάλισης προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι ένα θέμα που σηκώνει πολλή συζήτηση όπως φαίνεται εξάλλου. Εκεί που νομίζω όμως ότι πρέπει να είμαστε απόλυτοι και που δεν σηκώνει καμία έκπτωση είναι στην διασφάλιση της υγείας αυτών που θα υποστούν τους ελέγχους από τα συστήματα των body scanners. Ε, είμαστε απόλυτα βέβαιοι ή θα πειραματιζόμαστε. Και εμείς είμαστε μία από τις ομάδες εξάλλου ε, τη συχνή χρήση των αεροδρομίων, άρα είμαστε και μία από τι ομάδε των πειραματοζώων, εάν δεν είμαστε απόλυτα, απόλυτα βέβαια για τη διασφάλιση υγεία αυτών που θα χρησιμοποιούν τα body scanners. Ε, το δεύτερο ζήτημα είναι το κόστο, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επιβαρύνει τους ε, επιβάτε και το σύνολο των παραπάνω ερωτημάτων ε, τίθεται προσυζήτηση συζήτηση αν έχουμε την απόλυτη βεβαιότητα τη αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος. Διότι αν δεν είμαστε βέβαιοι ότι ε, είναι αποτελεσματικά στην, ε, για τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να τα υιοθετήσουμε, νομίζω ότι δεν σηκώνει ε, να συζητάμε ακόμα παραπέρα αυτό το θέμα. Ε, τέλος, είμαι από εκείνους που πιστεύουν στην υιοθέτηση ενός ενιαίου συστήματος εφαρμογής κανόνων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριος Μπράδμπορ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάνω δύο παρατηρήσεις θέλω μόνο. Οι συνάδελφοι νομίζω το ανέφεραν Βλέποντα τα ζητήματα αυτά, ιδιαίτερα σε σχέση με του ορατέ σώματο, τείνουμε να σκεφτούμε ότι κατά κάποιο τρόπο θα είναι η πανάκια για κάθε είδου ε, απειλή τρομοκρατική που αντιμετωπίζουμε. Στην πραγματικότητα όμω, αν το δούμε πιο ψύχρεμα, οι σαρωτέ σώματο ή οποιοδήποτε άλλο σαρωτή που βλέπουμε είναι μια τριτογενή, αν θέλετε, ε, μέθοδο για, να, ε, για να αποτραπούν άνθρωποι να επιβιβαστούν που φέρουν κάποιε συσκευέ. Πολλά από όσα χρειάζονται σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την προστασία των ε, επιβατών ουσιαστικά έχουν να κάνουν με συλλογή πληροφοριών και την παροχή, αν θέλετε, εκ των προτέρων προηγμένων πληροφοριών σε ό,τι αφορά του επιβάτε. ώστε να έχουν τα σχετικά συστήματα πληροφορίας, ε, να έχουν φορτωμένα τα στοιχεία σε ό,τι αφορά τα μοντέλα ε, ταξιδιού ε, των επιβατών κλπ. Αυτό μα ενδιαφέρει. Αν δούμε τα γεγονότα τη περασμένη εβδομάδα με τα εμπορεύματα, ουσιαστικά το γεγονό ότι καταφέραμε να προλάβουμε κάποια γεγονότα ήταν ακριβώ λόγω τη συλλογή πληροφοριών, όχι λόγω κάποιου ψαρωτή. Πρέπει λοιπόν να τα βάλουμε τα πράγματα σε κάποιο πλαίσιο όλο αυτού του μείγματο, αν θέλετε, όταν μιλάμε ευρύτερα για το θέμα τη ασφάλεια. Και πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά του ορατέ σώματο, η κυρία Φώστερ και άλλοι συνάδελφοι ήδη το ανέφεραν και συμφωνώ μαζί του θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς και προσεκτικοί, ώστε όχι απλώς σε ό,τι αφορά τους κινδύνους στην διασφάλιση απορρίτου και των ιδιωτικών στοιχείων, αλλά και τα θέματα διακύβευσης υγείας. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι κάποια από τα εφιστάμενα μοντέλα ε, σαρωτών στην αγορά είναι ασφαλή για τακτική χρήση. Η κυρία Φώστερ πολύ, πολύ συχνά, ε, πολύ σωστά εντόπισε το προσωπικό το οποίο μπαινοβγαίνει από τους σαρωτές αυτού στα αεροδρόμια. Ένας από τους συναδέλφους που είναι γιατρό, είπε ότι πραγματικά θα είναι ιδιαίτερη ιδιαίτερα σκεπτικός για την χρήση ενός σαρωτή ε, ακριβώς της υφιστάμενης, ε, ε της υφιστάμενης ε, μεθοδολογίας, της υφιστάμενης τεχνολογίας που υπάρχει, λόγω του ενδυνάμει κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος. Υπάρχουν πολλές σχετικά ανεκδοτολογικές ιστορίες, αλλά πρέπει να είμαστε απόλυτα πεπισμένοι και διασφαλισμένοι σε ό,τι αφορά τους κινδύνους υγείας για τα μηχανήματα, πρωτού συμφωνήσουμε για τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Το λέω γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν καλύψει τα θέματα που ήθελα να πω, γι' αυτό και δεν επεκτείνομαι. Πάντω, σίγουρα και τονίζω, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτή, αν θέλετε, την ευκαιρία σαν μια αντίδραση, αν θέλετε, σπασμωδική. Θα πρέπει να υπάρχει μια γενική ολιστική προσέγγιση και στρατηγική. Θα πρέπει να είμαστε προληπτικοί στη στρατηγική που εφαρμόζουμε σε κοινοτικό επίπεδο και όχι εκ των υστέρων βράτοντε. Ευχαριστούμε. Κύριε Κουμτσάκος, επόμενος. Τρία λεπτά. Ε, κύριε Πρόεδρε, η, η συζήτηση γίνεται στη βάση και στην υπόθεση ότι οι σαρωτές σώματος είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο. Διότι αν δεν είναι αποτελεσματικό, η συζήτηση που κάνουμε σήμερα πρέπει να πούμε ότι δεν έχει βάση. Θίγουμε με τη σημερινή συζήτηση την καρδιά μιας μεγάλης, ενός μεγάλου προβληματισμού πού βρίσκεται η ισορροπία μεταξύ αποτελεσματικής ασφάλειας και σεβασμού ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό η συζήτηση είναι δύσκολη, γι' αυτό εκφράζονται προβληματισμοί, γι' αυτό εκφράζονται ανησυχίες, ακόμα και μεγάλες επιφυλάξεις, αν όχι και αρνήσεις. Αλλά αυτή την μακρά συζήτηση οφείλουμε να την κάνουμε. Γιατί αν δεν την κάνουμε, αν δεν κάνουμε μια συζήτηση που αφορά την ποιότητα της δημοκρατίας μας, θα έχουμε δικαιώσει τους αντιπάλους της. Διότι θα έχουν καταφέρει το στόχο τους, δηλαδή να λιώσουν και να παραμορφώσουν το ίδιο το πολίτευμα το οποίο θέλουμε εμείς να προστατεύσουμε. Να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ των ρυθμίσεων σε ευρωπαϊκό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Υπάρχουν τρία ζητήματα που αλληλεξαρτώνται. Προστασία υγείας και τεχνολογία. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί δεν θα δημιουργεί προβλήματα υγείας. Προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων ιδιωτικής σφαίρας και ελέγχου των δεδομένων. Εδώ έχουμε δύο προκλήσεις. Πρώτον, να ελέγχουμε αποτελεσματικά και να προστατεύουμε αυτά τα δεδομένα και δεύτερον, αν θέλετε και μεγαλύτερη πρόκληση, είναι να πείσουμε τους πολίτες ότι είναι 100% σίγουροι ότι αυτά τα δεδομένα δεν θα, δεν θα αξιοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο. Άλλο είναι τι θα κάνουμε εμείς και δεύτερον είναι πώς θα πείσουμε ότι κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να τους προστατεύσουμε. Τέλος, για τον έλεγχο. Θα περνάνε όλοι ή θα υπάρχουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Εάν περάσουμε στην δειγματοληπτικό έλεγχο των επιβατών, εγείρονται άλλα ζητήματα. Με ποια κριτήρια θα γίνεται ο δειγματοληπτικό έλεγχο, με την εθνικότητα, με το χρώμα, με το πρόσωπο, με το πώ είναι ντυμένοι οι επιβάτε. Και εκεί είναι ζητήματα τα οποία, όπω σα είπα, θίγουν πολύ λεπτά, ε, πολύ λεπτά ζητήματα. Τέλο, κόστο. Η ασφάλεια είναι ένα δημόσιο αγαθό. Και επειδή είναι δημόσιο αγαθό, όλοι πρέπει να συμβάλλουν. Πιστεύω λοιπόν ότι και τα κράτη πρέπει να συμβάλλουν σε μεγαλύτερο ποσοστό και οι εταιρείε και τα αεροδρόμια. Και τελευταίοι σε αυτή την κλίμακα οι επιβάτες. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε μία λύση που να κατανέμει και να δίνει το κόστος μόνο σε έναν από αυτούς τους παράγοντες. Γιατί όπως σας είπα η ασφάλεια είναι δημόσιο αγαθό. Τέλος, όσον αφορά τους αρωτές εμπορευμάτων, εκεί δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα λεπτά ζητήματα και νομίζω ότι εκεί μπορούμε να προχωρήσουμε μεγαλύτερη ταχύτητα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ, Λάικφριντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα με επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω τον κύριο Λάγκενστάιν για αυτό που είπε και να πω, να επισημάνω κάτι σύντομο για το θέμα. Η κατάσταση όσα έχει δείχνει ότι κάποια κράτη-μέλη θέλουν να εισάγουν τους ε, σαρωτές, άλλοι όχι και νομίζω ότι η επίλυση της παρούσας κατάστασης είναι για μας να διασφαλίσουμε ότι αυτοί που θέλουν να εισάγουν τους αρωτές να το πράξουν σε συνθήκες όμως που θα είναι αποδεκτές σε όλους τους ανεξαρτήτους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτή είναι η δουλειά μας εδώ και το μέλημά μας. Όταν εξετάζουμε το θέμα σαρωτών σώματος πρέπει να ληφθούν πάρα πολλά πράγματα υπόψη. Όλα έχουν αναφερθεί από άλλους συναδέλφους, δεν χρειάζεται να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Το δεύτερο που είναι σημαντικό στην έκθεση αυτή είναι ότι δεν πρόκειται απλώς περί σαρωτών. Είναι μια έκθεση η οποία ασχολείται και με θέματα ασφάλειας στις ε, ΑΕΣ μεταφορές και είναι πολύ πιο σημαντική από την όλη συζήτηση περί σαρωτών, όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Μπράντον. Υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Χρησιμοποιώντα απλώ τεχνολογία δεν είναι ένα τρόπο επίλυση των πραγμάτων, θα πρέπει να είναι ένα συνδυασμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε και το θέμα του κόστου θα αντιμετωπιστεί και να μην επιβληθεί, αν θέλετε, στους ε, ταξιδιώτες, είναι δημόσια υποχρέωση και θα πρέπει να διασφαλιστεί από τις δημόσιες αρχές αλλά λόγω της προηγούμενης συλλογής πληροφοριών. Επομένως, θα πρέπει το θέμα της ασφάλειας των ε, αεροδρομίων να εκλειφθεί ως ένα σύνολο ανθρώπινων και τεχνικών παραγόντων. Εάν αφήσουμε ανοιχτή τη λάθος πόρτη σε λάθος ε, σημείο, ό,τι σαρωτή και να έχουμε, δεν πρόκειται να εξυπηρετήσει τίποτα. Άρα αυτή η διαδικασία που είναι μεικτή συνδυασμού, αν θέλετε, του ανθρώπινου παράγοντα και τεχνικών στοιχείων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα, η δική μας εργασία είναι αυτή του να θέσουμε όλες τις διαδικασίες ε, και τα πλαίσια για τη διασφάλιση, για την απόλυτη ασφάλεια στα αεροδρόμια ή πρέπει να γνωμοδοτήσουμε πάνω σε κάποιες τεχνολογίες οι οποίες εφαρμόζονται ενώ αφήκνονται πάνω σε θέματα υγείας, αποτελεσματικότητας στην ασφάλεια, σεβασμού των ε, προσωπικών και πολιτικών ελευθεριών και που δεν είναι να μην στεγογραφήσουμε, αν θέλετε, υποχρεωτικές τεχνολογίες. Θέλω να επιμείνω συγκεκριμένα σε κάποιες τεχνολογίες που είναι, αν θέλετε, ε, αποσκευές, ε, οι οποίες είναι, που κατεβαίνουν, αν θέλετε, που περνάνε χειραποσκευές, οι οποίες περνούν όμως μέσα από τα μηχανήματα ανείχνευσης. Γιατί αυτή τη στιγμή τελείως τεχαία κάνουμε δειγματοληπτικό έλεγχο μεταξύ 5 και 10% των αποσκευών ένας, ε, αν θέλετε, τρομοκράτης που είναι σε, σε αποστολή, αν θέλετε, σε αποστολή αυτοκτονίας, μπορεί κάλλιστα να περάσει την αποσκευή του μέσα από κανονικά τον ημάντα και δεν ενδιαφέρει. Το θέμα των στρατών, λοιπόν, το οποίο τίθεται, είναι το θέμα των ημάντων, αν θέλετε, που κινούνται ή δεν κινούνται προς τους άρωτες. Εάν κάνουμε σάρος του συνόλου των αποσκευών και είχαμε τα μέσα για κάτι τέτοιο, που θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρό, θα πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να κλείσουμε, θα πρέπει να κλείνουμε την ε, ε, επιβίβαση, αν θέλετε την καταγραφή των ε, αποσκευών, τρεις ώρες πριν από την αναχώρηση. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Δηλαδή ουσιαστικά θα εξαφανιστεί, το, θα εξαφανιστεί η αλληλογραφία το, του κατεπήγοντος, αν θέλετε, που θα πρέπει να γίνεται να διαβιβάζεται στο κατεπήγον. Σας υπενθυμίζω κύριε Πρόεδρε ότι οι αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από την Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα υγρά ήταν πραγματικά βιαστικές. Γιατί ξέρουμε πλέον ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε εγκαίρως τη σχετική ε, τεχνογνωσία για τη διασφάλιση ε, των υγρών προϊόντων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούν. Ο κύριος Κούν. Äh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι τελειοποιούμε την ασφάλεια της μετακίνησης των επιβατών, αλλά υπάρχουν κενά σε ό,τι αφορά τα εμπορεύματα, όπως είπαμε την περασμένη εβδομάδα. Για τις εμπορευματικές μεταφορές είναι υπεύθυνε οι εταιρείε, οι οποίες πρέπει να ανοιχνεύσουν τα εμπορεύματα, κάτι που είναι καθοριστική σημασίας για την Ευρώπη. Και αρμόδιες ε, αρχές ελέγχου λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα. Στη Γερμανία έχουμε μια αρμόδια υπηρεσία για τα, ε, τους επιβάτες που είναι η Ομοσπονδιακή Αστυνομία και αυτό είναι σημαντικό. δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε μετακινήσεις επιβατών αλλά και εμπορευματικές μεταφορές. υπάρχουν ε, μεταφορείς, ιδιωτικές ε, εταιρείε ε, οι οποίες είναι πιστοποιημένες και ελέγχουμε, ελέγχουμε συστηματικά κατά πόσο λειτουργούν με ασφαλή τρόπο. Στο αεροδρόμιο Σαλντεγκόλ τα εμπορεύματα ελέγχονται άμεσα με σκυλιά που θα μυρίσουν ε, εκρηκτικά και με άλλες διαδικασίες. Οπωσδήποτε ε, πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι των επιβατών, αλλά υπάρχουν και σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των εμπορευμάτων. Ταξίδεψα με την Air Berlin από το Αμβούργο στη Βαρκελόνη. Μου είπαν ότι εκεί υπήρχε ένας σαρωτής. Δεν είχα την επιλογή ε, να περάσω ή να μην περάσω. Και βρέθηκα ενώπιον του σαρωτή χωρίς να μπορώ να κάνω πίσω. Είδα λοιπόν τι συμβαίνει. Είδα ότι καταρχήν ε, έπρεπε να ακολουθήσουν τις οδηγίες οι χειριστές γιατί ήταν κάτι το καινούριο για αυτούς. Ε, έπρεπε να παραμείνω τρία δευτερόλεπτα με τα χέρια ψηλά και έπρεπε στη συνέχεια να περιμένω μερικά λεπτά, ίσως ένα λεπτό, έτσι ώστε να μου δώσουν το ok να περάσω μέχρι να προλάβει ο χειριστής να δει τη συνολική εικόνα. Ίσως τη βλέπουν και κάπου αλλού που δεν έβλεπα εγώ. Αλλά θα πρέπει να, να περιμένει κανείς ε, κάποιο χρόνο πριν του δοθεί το OK. Επίσης υπάρχει το θέμα ότι πρέπει να ε, βγάλουμε τα παπούτσια σε αυτήν την περίπτωση. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να περάσει κανείς από τον σαρωτή με τα παπούτσια. Επίσης ε, ο χειριστή, το χειριστή δεν τον βλέπουμε στην αρχή, τον βλέπουμε στο τέλος της διαδικασίας. Αυτή ήταν η προσωπική μου εμπειρία. Άρα μπόρεσα να φτάσω σε ορισμένα συμπεράσματα. Εάν μπορούμε να δεχτούμε το συνολικό κόστος ως προς την ασφάλεια, ως προς το χρονικό καθαρά σε σχέση με αυτό που κερδίζουμε στην ασφάλεια, τότε θα μπορούσα να το δεχτώ, γιατί σίγουρα κερδίζουμε στην ασφάλεια και ας χάνουμε χρόνο. Θα πρέπει να δούμε όμως ε, πώς θα έχει το συνολικό κόστος και έτσι το θέμα των φορτίων και των ε, υγρών θα το δούμε αργότερα. Ιδιαίτερα ως προς τα υγρά τα οποία θα αποφασίσουμε εάν περνάνε από σαρωτές ή όχι. Βεβαίως ένας απαράβατος όρος είναι η υγεία. Είπαμε γυναίκες, έγκυες γυναίκες, παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να ακολουθούν μία άλλη διαδικασία. Αυτό αφορά και τους τακτικούς επιβάτες και τους χειριστές, δηλαδή να δούμε κατά πόσο υπάρχει επίπτωση στην υγεία τους. Και βεβαίως το θέμα της ιδιωτικότητας είναι ένα σημαντικό θέμα, δηλαδή οι εικόνες θα πρέπει να καταστρέφονται αμέσω. Ευχαριστώ και πολύ σύντομα. έχουμε νομίζω καταλήξει σε ορισμένες πρακτικές σε αυτό τον τομέα. Αλλά υπάρχουν και τα μικρά αεροδρόμια Ορισμένοι από εσά έχουν δει σαρωτέ σώματος, άλλοι όχι. Υπάρχουν λοιπόν διαφορές από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο και από χώρα σε χώρα, όπω διαπιστώσαμε και από τη συζήτηση που είχαμε εδώ. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στα μεγάλα αεροδρόμια και στα μικρά αεροδρόμια. Στα μεγάλα αεροδρόμια υπάρχουν συστήματα ασφάλειας, αλλά στα μικρά δεν ξέρω τι γίνεται. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Ίσως θα μπορούσε να έρθει κάποιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, ίσως θα μπορούσαμε να φέρουμε ορισμένου ανθρώπους που εργάζονται στα μικρά και στα μεγάλα αεροδρόμια για να μας πούν ακριβώς τι συμβαίνει. Ένα μικρό αεροδρόμιο είναι πάρα πολύ δύσκολο να εγκαταστήσει ε, σαρωτές σώματος, δεν υπάρχει επαρκής χώρος. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε επιτόπου για να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται. Αυτό προτείνω. Ευχαριστώ. Προτού δώσω το λόγο για θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεγκράντες Πασκουάλ για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα που και η έκθεσή του θα είναι ασφαλώς πολύ λεπτομερής. Επανέρχομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Μπακμπορν. Εάν στηριχθούμε, αν περιμένουμε ότι θα, ανακαλύψουν τους τρομοκράτες τα αεροδρόμια, είμαστε καταδικασμένοι σε αποτυχία. Διότι δεν είναι δουλειά των αεροδρομίων να ανακαλύπτουν τους τρομοκράτες. Το αεροδρόμιο είναι τελευταία γραμμή ε, άμυνας. Και αυτό πρέπει να καταστεί από την αρχή απόλυτα σαφές. Σχετικά με τα εμπαρεύματα μέχρι ποιου σημείου στην ε, ε, αλυσίδα θα φτάσουμε. Σε όλα τα κέντρα διανομής θα πάμε και θα τους πούμε ότι εκείνοι πρέπει να εγκαταστήσουν σε ρωτή διότι υπάρχει μια ολόκληρη αλυσίδα για τις ε, εμπορευματομεταφορές. Και αν στηριχθούμε μόνο στα αεροδρόμια, και πάλι είμαστε καταδικασμένοι σε επιτυχίες, σε αποτυχία. Αν οι Αμερικανοί λένε κάτι, υπάρχουν κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιδρούν απλά και μόνο επειδή το, το είπαν οι Αμερικάνοι. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την ε, ε, αντίδραση. Και σχετικά με τον body scanner, είναι παραμύθι ότι είναι εθελοντική η χρήση του. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, αν αρνηθείτε να περάσετε από τον body scanner, απλά και μόνο δεν θα ταξιδέψετε, δεν θα πετάξετε. Δεν είναι λοιπόν εθελοντική η χρήση του. Υπάρχουν ασυνέπειες και διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Αλλά στο εσωτερικό των κρατών μελών, το Heathrow στο Heathrow ή στο Τελαβίβ περνάει κανείς από πάρα πολύ αυστηρούς ελέγχους. Σε άλλα αεροδρόμια η έλεγχη είναι τελείως διαφορετική. Πολύ λιγότερο συστηματική και πολύ λιγότερο εκτεταμένη. Και αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε αυτές οι ασυνέπειες, αυτές οι ασυνέπειες που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες χώρες και ανάμεσα στα διάφορα αεροδρόμια. Και να σας πω και κάτι, οι Ηνωμένε Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται, δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την υιοθέτηση μιας ενιαίας λύσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόβλημα είναι αυτό και ως ότου λύσουμε αυτό το πρόβλημα και προωθήσουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την... Ε, θα συνεχιστεί εσαΐ αυτή η συζήτηση και όταν οι τρομοκράτες το διαπιστώσουν αυτό αφού θα μόλις επιτεθούν ε, για μια φορά ε, σε ένα τρένο, τότε θα, καθιερώσουμε, θα, καθιερωθούν, θα καθιερωθούν σε ορισμένα κράτη-μέλη ή σαρωτέ σώματος και για τους σιδηροδρόμους, επειδή το απαιτούν αυτό οι Ηνωμένε Πολιτείε. Πρέπει λοιπόν να γνωρίσουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε, να συσπηρωθούμε συνάδελφοι και να προωθήσουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ώστε να μην κινείται ο καθένας με το δικό του τρόπο. Ο κύριος Καλιάκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Δεγκράντες για την ε, πολύ καλή παρουσίασή του και όλα τα μέλη επίσης που συμμετέχουν στη συζήτηση. Νομίζω ότι όλα τα θέματα έχουν τεθεί επιτάπτως και νομίζω ότι όλοι συμφωνήσαμε ε, για τη σημασία ενίσχυσης της ασφάλειας και τη σημασία του να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες μας θα προστατεύονται. Και υπό αυτή την έννοια θα ήθελα να πω εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και της Γενικής Διεύθυνση Αεροπλοεία από την 11η Σεπτεμβρίου οι αεροπορικές μεταφορές είναι αναπόσπαστο κομμάτι ασφάλεια σε ό,τι αφορά τη σχετική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντοπίσαμε την εποχή εκείνη τον μεγάλο αντίκτυπο των τρομοκρατικών ενεργειών στο σύστημα αεροπλοείας και έκτοτε η αεροπλοεία είναι πάντα υπό απειλή. Υπήρξαν πάρα πολλές απόπειρες έκτοτε. Είχαμε ε, βομβιστές, ε, ε, είχαμε τα υγρά εκρηκτικά υγρά στο Χήθρο. Είχαμε την, ε, το γεγονός ε, το συμβάν του Σεπτεμβρίου και τις πρόσφατες ε, απόπειρες με τη μεταφορά εκρηκτικών δεμάτων. Είμαι κάπως λιγότερο απεσιόδοξο από τους άλλους ομιλητές. Στην Ευρώπη έχουμε κοινούς κανόνες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της αεροπλοείας που εγκρίθηκαν χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε χρόνο ρεκόρ μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Έχουμε τον κανονισμό 2320 του 2002 που ήταν η άμεση αντίδραση αλλά βελτιωθήκαμε έκτοτε και συνεχώς παρακολουθούμε την κατάσταση. Το τελευταίο παράδειγμα είναι ο κανονισμός 300 του 2008 που επίσης βελτίωσε και ενίσχυσε το σύστημά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πολύ ισχυρό και εύρωστο σύστημα που καλύπτει και τους επιβάτες και τα εμπορεύματα και που διασφαλίζει ότι λειτουργεί η εσωτερική μας αγορά, αλλά που επίσης διασφαλίζει ότι έχουμε ευρωπαϊκά πρότυπα και κανόνες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που, εφαρμόζονται από κοινού και ενιαία. Ετέθη από τον κύριο Γκράντε ένα ερώτημα από την αρχή. Κατά πόσον η έκθεσή του θα έπαιρνα καλύπτει μόνο τους αρωτές ασφαλείας ή και άλλα ζητήματα. Νομίζω ότι η συζήτηση κατέδειξε ότι είναι πολύ σημαντικό να καλυφθούν και άλλα ζητήματα που άπτονται τα θέματα ανασφαλείας και θα ήθελα να αναφέρω τέσσερα πολύ σημαντικά. Πρώτον, ε, οι σαρωτές ασφαλείας και θα αναφέρω στην Επιτροπή που βρισκόμαστε σχετικά. Δεύτερον, θέματα εμπορευμάτων και θα αναφέρω επίσης και θα δώσω στην Επιτροπή κάποιες προφορίες σχετικά. Νομίζω όμως ότι ο κύριος Κάλλας, ο οποίος θα έρθει σε κανένα δεκάλεπτο, πιθανότητα θα παράσχει επιπρόσθετα στοιχεία στην Επιτροπή. Νομίζω ότι θα πρέπει να αγνοήσουμε και τη διεθνή διάσταση του θέματος και τέλος έχουμε και τα θέματα χρηματοδότησης. Ας ε, ξεκινήσω με το πρώτο θέμα, τους αρωτέ ασφαλείας. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του θέματο αυτού. Όλες οι παρεμβάσεις ε, υπογράμμισαν τη σημασία του να υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση. Η ενισχύη κατάσταση είναι το απόλυτο κατακαιρματισμό. Κάποιες χώρες ε, είναι σε φάση ελέγχου, σαρωτών ελέγχου. Το κάνουν με βάση ε, ε, ελέγχου στο Σίπολ, στο Ελσίνκι, στο Χίθρο, στο Μάντσεστερ, σε κάποια αεροδρόμια τέλο πάντων. Και γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν κοινοτικοί κανόνε επί του θέματο αυτού. Το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να υπάρξουν, να θεσπιστούν σχετικοί κοινοί κανόνε. Και άκουσα τη σχετική κριτική, την οποία ανακλαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά πιθανότατα δεν είχαμε διεξοδικά σκεφτεί, σκεφτεί το θέμα. Ίσως ε, να, ε, να δράσαμε, αν θέλετε, πολύ πρόωρα και το σκεφτήκαμε και επανήλθαμε και υποβάλαμε αυτή την έκθεση τώρα για να λάβουμε τις απόψεις σας, να δούμε ποια είναι τα σημεία κλειδιά που θα θέλετε να αντιμετωπίσουμε στο θέμα. Τώρα κάνουμε μια ε, αξιολόγηση του αντίκτυπου του ε, νομοθετήματος αυτού και που θα καλύψει όλα τα θέματα που αναφέρετε. Θα ασχοληθεί με τα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, θα ασχοληθεί με τα θέματα υγείας, θα ασχοληθεί με τα θέματα ιδιωτικότητας και θα ασχοληθεί και με τα θέματα κόστους. Και θα υπάρξουν αρκετές εναλλακτικέ που θα υποβληθούν. Θέλουμε να συνεχίσει η παρούσα κατάσταση. Θέλουμε τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν με δοκιμές και, όλο, και την υιοθέτηση όλο και πιο αυστηρών μέτρων. Θέλουμε να επιβάλλουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεωτικά τους αρωτές ασφαλείας θα πρέπει να υπάρχει μια εναλλακτική για χώρες που πιστεύουν ότι υπάρχει την πιθανότητα αυτή να τους έχουν και να τους άγουν. Υπό ποιες συνθήκες. Νομίζω ότι όλα τα ερωτήματα είναι θεμητά και έχουν τεθεί επιτάπτως και τα οποία αυτή τη στιγμή είναι υπό εξέτωση από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε επίση διαβουλευτεί με την Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και επίσης βρισκόμαστε στη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους και τις σχετικές υπηρεσίες ακούσαμε, είχαμε μια σειρά εκροάσεων και μόλις πρόσφατα λάβαμε σχετικές προφορίες. Είμαστε αρκετά προωθημένοι σχετική δική μας εργασία και ελπίζουμε ότι του χρόνου θα μπορούμε να υποβάλουμε αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ποιε εναλλακτικέ είναι στη διάθεσή μα. Και προτού υποβάλουμε προτάσει, θα θέλαμε να προηγηθεί συζήτηση. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν λύσει. Εξαρτάται όμω εν πολλής από το πόσο θέλουμε να προχωρήσουμε στο πεδίο αυτό. Τα κράτη-μέλη πιστεύουν ότι οι σαρωτές ασφαλείας έχουν προστιθέμενη αξία και μπορούν να προσφέρουν στην ανείχνευση μη μεταλλικών επικίνδυνων αντικειμένων και γι' αυτό και χρησιμοποιούνται. Είναι επίσης ε, δυνατό, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν διεξαχθεί, να αντιμετωπιστούν τα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδιωτικότητας, αλλά και τα θέματα υγείας θα θέλαμε όμω όταν έρθουμε στο Κοινοβούλιο, αφήσει να έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη αυτή των επιπτώσεων, να συζητήσουμε τις αλλακτικέ που έχουν στη διάθεσή μα. Τώρα, για τα εμπορεύματα. Πάρα πολλά θέματα αναφέρθηκαν σχετικά. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι εναρμονισμένοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τα εμπορεύματα υπάρχουν από το 2003. Το 2010 εισήχθη ένα νέο πακέτο νομοθετικών μέτρων για την ασφάλεια τη αεροπλοεία. Το σύστημα βασίζεται σε δύο πυλώνε. Ασφάλεια τη εφοδιαστική αλασίδας, όπω αναφέρθηκε, και η των εμπορευμάτων, των αποστολών. Και παρακολουθούμε συνεχώ την εφαρμογή όλων των σχετικών κανόνων ασφαλείας τη αεροπλοεία που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βοηθούμε επίση τα κράτη-μέλη για την σωστή εφαρμογή και κάτι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αναφέρθηκε από πολλού ομιλητέ και του ευχαριστώ που έθιξαν το ζήτημα πρέπει να κάνουμε περισσότερο στο πεδίο της έρευνας. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές δυνατότητες. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν σημαντικοί τρόποι εργασίας που πιθανότατα δεν αντιμετωπίζουμε τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε στο πεδίο της έρευνας και ανάπτυξης. Και υπάρχουν δυνατότητες ενίσχυσης του θέματος αυτού. Και είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε και με του ειδήμονε, του εμπειρογνώμων την περασμένη Παρασκευή. Την περασμένη Παρασκευή συνήλθε σε έκτακτη συνάντηση η Επιτροπή Εμπειρογνωμών ασφαλεία Αεροπλοεία και τέθησαν τέσσερα πολύ σημαντικά σημεία στα οποία συμφώνησαν. Πρώτον, χρειαζόμαστε σε σχέση με τα εμπορεύματα να χρησιμοποιήσουμε μια προσέγγιση επί τη βάση αποτίμηση κινδύνου, λαμβάνοντα υπόψη την ποιότητα τη άρρωση, την δρομολόγηση, την φύση των αποστολών και τον τύπο ε, πτήσεων που μεταφέρονται συγκεκριμένα εμπορεύματα. Η Ευρώπη έχει 10 από του 20 κορυφαίου ε, κόμβου τη Ευρώπη. Το 20% όμως των εμπορευμάτων μετακινούνται με ε, επιβατηγές πτήσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν να το εξετάσουμε το θέμα αυτό και να αποφασίσουμε τους τρόπους για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Δεύτερο σημείο πολύ σημαντικό, η διεθνής διάσταση, η οποία τονίστηκε από πολλούς ε, ομιλητές. Πρέπει να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ, αναφέρθηκε αυτό, αλλά όχι μόνο με τις ΗΠΑ, η αεροπλοεία είναι παγκόσμια. Έχουμε τον ΙΚΑΟ, το Διεθνή Οργανισμό ε, Αεροπλοεία. Στη Γενική του Συνέλευση υπάρχει πολύ σημαντική ατζέντα για συνεργασία και πρέπει να αναπτύξουμε με διεθνεί εταίρους πολύ σημαντικές σχετικέ δραστηριότητε. Είναι θεμελιώδε να εργαστούμε για την ανάπτυξη των ικανοτήτων. Υπάρχουν ζητήματα σε τρίτες χώρες που χρήζουν αρρωγίες για να αναπτύξουν το δυναμικό τους. Αλλά γενικά χρειαζόμαστε παγκόσμια πρότυπα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να ενισχύσει τις εκθεωρήσεις ώστε να επιτύχει πλήρη και σωστή εφαρμογή των κανόνων και να εφαρμόσει σημαντικές και γενοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες για την σάρωση. Σε σχέση τώρα συγκεκριμένα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, του χρόνου θα έχουμε στην Ουάσιγκτον την Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΕ. Δεν είναι μια μυστική επιτροπή, συμμετέχουν οι βιομηχανίες και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις του Διατλαντική ε, αγοράς αεροπλοείας, γιατί τα κράτη-μέλη πλέον δεν έχουν διμερείς συμφωνίες με τι ΗΠΑ οι οποίες συμφωνίες γίνεται μέσω της ανοιχτή συμφωνία Ανοιχτών Εθέρων Ευρωπαϊκής Ένωση ΕΠΑ. Έχουμε σημαντικά ζητήματα προ συζήτηση και ήδη παρέχουμε τακτικά στην Επιτροπή Μεταφορών όλες τι απαραίτητε πληροφορίε. Είναι μια τεχνική συζήτηση, αλλά είναι σημαντικό να είναι ενήμερο το Κοινοβούλιο επί των εξελίξεων στο πεδίο αυτό και σημειώνουμε πρόοδο δεν έχουμε τους ίδιους κανόνες από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ίσως κάποια στιγμή φτάσουμε σε κοινή συμφωνία. Αλλά πάντως η θέση μας δεν είναι να εφαρμόσουμε τα αμερικανικά πρότυπα. Σε κάποια ζητήματα δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι. Θέλαμε εμείς να κάνουμε περισσότερο. Είναι ένας διάλογος μεταξύ εμπειρογνωμόνων, όπου εν κατακλείδη αυτό που θέλουμε εμείς είναι να αξιολογήσουμε την ισοτιμία, ώστε να έχουμε ενιαία ασφάλεια που θα διευκολύνει την ε, ε, μετακίνηση των επιβατών. Τέλος, από πλευρά μας, θα ήθελα επίσης να επισημάνω και να ε, υπογραμμίσω τη σημασία της χρηματοδότησης. Υπάρχει σχετική πρόταση επί της οποίας έχει ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ένα θέμα βεβαίως που θα τεθεί με την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε ποιες είναι οι προοπτικές. Είναι πολύ μεγάλη ζήτηση για το ποιο πληρώνει. Πολύ σωστά επισημάθηκε από πολλού ομιλητέ και είναι στεμελιώδη ζήτημα. Εν κατακλείδη, η Ευρώπη προσβλέπει στην στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και προσβλέπουμε επίσης στην διευκόλυνση ώστε να χορηγηθούν όλες οι απαραίτητες προφορίες που ζητούνται και να συνεργαστούμε με τον κύριο Ντεγκράντες και τα μέλη των διαφόρων επιτροπών προκειμένου να έχουμε το πιο ισχυρό σύστημα ασφαλείας που θα μπορούσαμε να έχουμε, αλλά όπως ελέγχθη από πολλούς ομιλητές, εξασφαλίζοντας σωστή ισορροπία με τα ιδιωτικά συμφέροντα, με τα θεμελιώδη δικαιώματα, με τα θέματα ανθρώπινης υγείας, με όλα τα συμπαρομαρτούντα γιατί αν κατακλείδη θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη σημασία της αεροπλοείας για την κοινωνία μας και τη σημασία των αέριων μεταφορών για την οικονομική μας ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καγιάκο. Κύριε Ντεγκράντες, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Έχουμε λίγο χρόνο, αλλά να είστε όσο γίνεται πιο σύντομος. Βεβαίως έχετε δικαίωμα να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, χωρίς καμία εξαίρεση, αρχίζοντας από τον προλαλήσαντα, από την Κομισιόν δηλαδή. Μας ενδιαφέρει η μελέτη αντικτύπου. Όταν δημοσιευθεί, θα δούμε κατά πόσο μπορούν να επιληθούν τα προβλήματα που θέσαμε. Υπάρχει μια βασική συμφωνία από όσο κατάλαβα από όλους τους ομιλητές. Δεν θα περιοριστούμε μόνο στους ε, σαρωτές σώματος, αλλά θα ασχοληθούμε σφαιρικά με την ασφάλεια στην αεροπλοεία. Βεβαίως δεν μπορούμε να αναθεωρήσουμε όλα τα πλαίσια. Αυτό θα ήταν ε, τρέλα. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για όλες, ως προς όλες τις πτυχές της αεροπλοείας. Υπάρχει μεγαλύτερη συμφωνία από ό,τι φαίνεται. Πολλά θεμητά ζητήματα τέθησαν, τα οποία είναι παλαιά ζητήματα και ερωτήματα. Πρόκειται για ανησυχίες που είχαμε ήδη εκφράσει και η τεχνολογία έλυσε μερικές από αυτές. Βεβαίως υπάρχει η ανησυχία της υγείας, στο τομέα της υγείας. Δεν θα πρέπει να πλήτεται η υγεία από τις ε, τεχνικές λύσεις που βρίσκονται. Επίσης, ως προς την διατήρηση των στοιχείων, γιατί είναι σαφές ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό. Σε αυτό θα επιμείνουμε. Επίσης, οι νέες τεχνολογίες θα πρέπει να αποτελέσουν προστιθέμενη αξία και να δώσουν αναλογικότητα στην αντιμετώπιση των κινδύνων που όλο ένα και επαυξάνονται όπως γνωρίζουμε από την κοινωνική πραγματικότητα. Βεβαίως δεν πρέπει να αντιδρούμε απλώς, διότι η τρομοκρατία είναι μια καθημερινή διαδικασία. Οι τρομοκράτες προσπαθούν να πλήξουν τις δημοκρατικές ε, κοινωνίες. Γι' αυτό θα πρέπει βαθμιδών να εφαρμόσουμε συγκεκριμένα μέτρα. Βεβαίως θα πρέπει να προτρέξουμε έναντι της τρομοκρατίας. Και όπως είπε ο συνάδελφος Δίας Δεμέρα, δεν αντιμετωπίζουμε τις ίδιες ε, δυσκολίες ε, ως προς τους σαρωτές φορτίων. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα 50% των φορτίων μεταφέρεται ε, από τις ίδιες πτήσεις που μεταφέρουν και επιβάτες. Περνάνε βεβαίως ακτίνες, θα πρέπει να περνάνε ακτίνες χ. Μιλάμε λοιπόν για θεμελιώδη δικαιώματα που αφορούν τους σαρωτές σώματος. Εδώ θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα ιδιωτικότητας. Βεβαίως είναι ένα μέτρο το οποίο δεν μπορούμε να, δώσουμε, να δούμε απομονωμένα. Δεν θα πρέπει να πληγεί η εναέρια κυκλοφορία. Θα πρέπει να ελέγξουμε και τις χειραποσκευές βεβαίως. Να δούμε τι θα κάνουμε και με τα υγρά των χειραποσκευών. Έχουν ληφθεί αποφάσεις, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα αρκεστούμε σε αυτές. Θα προβάλλουμε μία συνολική αποστολή και βεβαίως χρειαζόμαστε χρόνο για όλα αυτά. Εγώ ασχολήθηκα με τους αρωτές σώματος, αλλά θα πρέπει να διευρύνουμε το θέμα όπως ζητήθηκε ομόφωνα έτσι ώστε να ασχοληθούμε ολοκληρωμένα με την ασφάλεια της αεροπλοείας. Γι' αυτό θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για αυτή τη συνολική προσέγγιση. Και βεβαίως θα πρέπει να μιλήσουμε με την Επιτροπή για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία της μελέτης αντικτύπου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στην προσέγγισή μας. Ευχαριστώ κύριε έγινε μια προκαταρκτική συζήτηση για τις, θα προβλέπετε μια προκαταρκτική συζήτηση για τις 5 Νοεμβρίου και αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεστε χρόνο για να διευρύνετε την κάλυψη του θέματος και περιμένουμε και τα αποτελέσματα και, και θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα αποτελέσματα της ε, αξιολόγησης των επιπτώσεων. Σχέδιο έκθεσης 25 Ιανουαρίου, ψηφοφορία Επιτροπή Μεταφορών γύρω στο Μάρτιο και η ψηφοφορία στη, στην Ολομέλεια το Μάιο του 2011. Αυτό που προέχει να γίνει η δουλειά σωστά και όχι βιαστικά. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσετε να τηρήσετε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ και όλα τα μέλη για την πειθαρχία τους, για το γεγονός ότι τήρησαν το χρόνο που τους είχε δοθεί, τους εκπροσώπους των άλλων επιτροπών για τη συμβολή τους σε μια, κατά την άποψή μου, πολύ καλή και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τώρα θα περιμένουμε την άφηξη του Επιτρόπου Κάλλας. Okay, colleagues, can Ο αντιπρόεδρος, ε, υποδεχόμαστε τον αντιπρόεδρο κύριε Κάλλες, έχουμε μια ώρα και 50 λεπτά και θα σας ζητήσω να είστε πειθαρχημένοι στις παρεμβάσεις σας και θα αρχίσουμε αμέσως με τον Επίτροπο. Κύριε Κάλλας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι το πρόγραμμα εργασίας και διαρθρωτικός διάλογος, αλλά βεβαίως θα είμαι ε, πρόθυμος να συζητήσω και το θέμα των αεροπορικών μεταφορών. Παρακαλώ όσους φεύγουν να φεύγουν χωρίς να κάνουν φασαρία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα εργασίας και μετά ας δούμε ενδεχομένω και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας για τα επόμενα χρόνια στις 27 Οκτωβρίου και είμαι πάντοτε πάρα πολύ ευτυχής που μου δίνετε ευκαιρία να το συζητήσω μαζί σας. Το πιο σημαντικό έγγραφο για το επόμενο χρόνο είναι η Λευκή Βίβλος για το μέλλον των μεταφορών που πρόκειται να παρουσιάσω στις αρχές του επόμενου έτους. Για να υπάρξει συνέπεια με τις άλλους τομείς πολιτικής στα πλαίσια της διαδικασίας Ευρώπη 2020, θα, η Λευκή Βίβλος θα υποβληθεί μαζί με άλλα σημαντικά κείμενα πολιτικής για τη θέμα της ενέργειας και του κλίματος. Θα προσπαθήσουμε να συγχωνεύσουμε ορισμένες σκέψεις και ορισμένες ιδέες για να έχουμε μια λευκή βίβλο η οποία θα αναφέρεται όχι μόνο σε συγκεκριμένου τομείς αλλά σε κοινέ προσπάθειες. Η λευκή βίβλο για τις μεταφορές θα στηριχθεί στους εξή πυλώνες. Εσωτερική αγορά, καινοτομία και υποδομές. Μια ανταλλαγή απόψε με τους Υπουργούς Μεταφορών οργανώθηκε στο τελευταίο Συμβούλιο Μεταφορών στις 15 Οκτωβρίου του 2010 που εστιάστηκε στις σημαντικότερες προκλήσεις για τις μεταφορές στο μέλλον και το ρόλο των νέων τεχνολογιών. Τα κράτη-μέλη υποστήριξαν μια βιώσιμη, αποτελεσματική και καινοτόμο πολιτική μεταφορών. Ωστόσο, υπήρξαν αποκλίνουσες απόψεις σχετικά με τις δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα οι απόψεις διέφεραν σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των πρόσθετων αναγκών σε θέματα υποδομής από τον κοινοτικό προπολογισμό. Το 2011 θα ε, ε, ξεκινήσει με την έναρξη των συζητήσεων για τη χρηματοδότηση και τα προγράμματα για το επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο και αυτό θα είναι το κλειδί για τον τομέα των μεταφορών ελπίσης. Οι, προπο... προτάσεις μας πρόκειται να επαυληθούν πριν από τις θερινές διακοπές και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα σας παρουσιάσω το πρόγραμμα εργασίας με βάση πέντε προτεραιότητες όπως διατυπώθηκε στην διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών στην επιστολή που έστειλαν τον Ιούλιο. Θα ξεκινήσουμε με την εσωτερική αγορά, ένα σημαντικό στοιχείο για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών. Πρώτα, ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς σε όλους σε όλα τα συστήματα μεταφορών. Πρόσφατα λάβατε την ε, αναμόρφωση ε, του πρώτου πακέτου, της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Ελπίζω θα συνεχιστούν οι συζητήσεις για τα δικαιώματα των επιβατών ε, λεωφορείων και πούλμαν και ότι θα υπάρξει, θα επιβληθούν αυστηρότερες χειρώσεις για τις κυκλοφοριακές παραβιάσεις θα παρουσιάσω μια ανακοίνωση για τα δικαιώματα των επιβατών που θα αξιολογεί τους ισχύοντες κανόνες που εφαρμόζονται για όλα τα μεταφορικά συστήματα. Κατόπιν το 2012 θα ακολουθήσει μια νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών της αεροπλοείας ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις ε, της ε, ε, ηφαιστειακής τέφρας που έγινε με την προϋπόθεση ότι τα, η αξιολόγηση των επιπτώσεων δείξει ότι υπάρχει ανάγκη για την αναθεώρησή της. Επίσης μελετούμε την ανάγκη ενίσχυσης των δικαιωμάτων των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης μια εταιρεία το οδικό καμποτάζ ε, εξακολουθεί να περιορίζεται και σκοπεύω να δημοσιεύσω μία έκθεση το 2012 για τη λειτουργία της, ε, της εσωτερικής αγοράς ε, οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Σε ό,τι αφορά τον τομέα των σιδηροδρόμων, μια ανακοίνωση για την η πρόσβαση στην, ε, αγορά, στη σιδηροδρομική αγορά του 2012 θα εξετάζει την οργάνωση της αγοράς αυτής συμπεριλαμβανομένων ε, του ανοίγματο της αγοράς για τις μεταφορές ε, χώρες μεταφορές επιβατών με βάση μια αναμόρφωση του της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Επίσης θα ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων το 2012. Τέλος, θα παρουσιάσω το 2011 ένα πακέτο για την ηλεκτρονική κινητικότητα, η mobility, που θα αναφέρεται στη χρήση τεχνολογίες από διάφορα συστήματα μεταφορών για καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και μεγαλύτερη ασφάλεια και ευρύτερη δυνατότητα επιλογής για τους καταναλωτές. Θα καλύπτει διάφορα θέματα, όπως μια πρόταση για οι ηλεκτρονικές θαλάσσιες μεταφορές, την αναμόρφωση της, του ψηφιακού ε, ταχογράφου, της νομοθεσίας για τους ψηφιακούς ταχογράφους για καλύτερη προστασία από απάτες και παραποίησεις, μια αναθεώρηση κατάστασης επίσης σε ό,τι αφορά τη χρήση ηλεκτρονικών διοδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάπτυξη των υποδομών και καινοτομία. Συμφωνώ με την Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι οι κατάλληλες ε, ε, υποδομές μεταφορών είναι μια από τις προτεραιότητές μας. Ετοιμάζουμε, προβαίνουμε τώρα σε μια αναθεώρηση των ε, κατευθυντηρίων γραμμών που ισχύουν για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών για το πρώτο εξάμεινο αυτού του έτους που θα συνοδευτεί από μια έκθεση για την εφαρμογή των των TEN-T, διευρωπαϊκών δικτύων ε, στον τομέα των μεταφορών. Για να προωθήσουμε την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών, ετοιμάζουμε επίσης ένα σχέδιο στρατηγικής ε, ένα στρατηγικό σχέδιο για την τεχνολογία των μεταφορών που θα καθιερώσει ένα στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη προκειμένου οι μεταφορές ε, να καταστούν πιο βιώσιμες μέχρι τον ορίζοντα τον χρονικό του 2050. Συνεργάζομαι με άλλους επιτρόπους για να ετοιμάσουμε μια ανακοίνωση για τη διεθνή πολιτική μεταφορών σχετικά με τις γειτονικές χώρες η προστασία του περιβάλλοντος. Για την, η καλύτερη, για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, σημαντικό το μέρος των μεταφορών να περιορίσει τις εξωτερικές του δαπάνες. Η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει μια αναθεώρηση της οδηγίας για την Οροβινιέτ που συζητούν αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Με ιδιαίτερη ευτυχή ότι το Συμβούλιο υποστηρίζει τα βασικά στοιχεία αυτή τη αναθεώρηση. Όταν εγκριθούν, θα καθιερώσουν την αρχή τη εσωτερικοποίηση των εξωτερικών δαπανών στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η Λευκή Βίβλο θα εξετάσει και άλλε περιβαλλοντικέ πτυχέ και ειδικότερα το σημαντικό θέμα της μείωσης των ε, εκπομπών άνθρακα και της ε, ε, διακοπής διακοπής της, εξάρτησης των μεταφορών από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό είναι μια, ε, κάτι που εκτείνεται πέρα, ε, καλά πέρα από την χρονική προοπτική του 2011 θα πάρει τη μορφή μιας ανακοίνωσης για καθαρά συστήματα μεταφορών με σχετικές νομοθετικές προτάσεις που θα γίνουν το 2012. Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει κοινωνικό διάλογο με διάφορα μεταφορικά μέσα για να προκειμένου να διευκολύνει τις συζητήσεις ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους. Η Λευκή Βίβλος θα συζητήσει τις κοινωνικές στοιχές της πολιτικής των μεταφορών. Σκοπεύω το 2011 να παρουσιάσω επίσης ένα πακέτο, μια δέσμη μέτρων για το, το πρόγραμμα των κοινωνικών θαλασσίων μεταφορών που στηρίζεται σε τρία στοιχεία. Μια ανακοίνωση για την κοινωνική ατζέντα των θαλασσίων μεταφορών, μια νομοθετική πρόταση για την ενίσχυση της σύμβασης του ILO και την αναθεώρηση της οδηγίας για την ε, <clears throat> εκπαίδευση των ναυτικών. Πέμπτον, ασφάλεια και ε, κατευθύνεται για την ασφάλεια και την προστασία και μετρήσιμη στόχοι για όλα τα μεταφορικά μέσα. Αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Για την ασφάλεια έχουμε πρόσφατα εγκρίνει την αναθεώρηση του κανονισμού για την ΕΜΣΑ, για την Ευρωπαϊκή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θαλάσσιας ε, Ασφάλειας του χρόνου, εκτός από το κοινωνικό ε, πακέτο για τις θαλάσσιες μεταφορές θα εξυγχρονίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την κοινοτική νομοθεσία για την ασφάλεια των επιβατών στα πλοία. Για την ασφάλεια θα αξιολογήσουμε την παρούσα κατάσταση συμπεριλαμβανομένων και των, των σημερινών και των μελλοντικών απειλών και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την χρήση των ε, ε, σαρωτών ασφαλείας που είναι ένα ευαίσθητο θέμα που προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον. Προσπάθησα λοιπόν να σας παρουσιάσω σύντομα τις βασικές προτεραιότητές μου που ταυτίζονται πάρα πολύ με αυτά που έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και να προσθέσω κάτι ακόμα για του χρόνου. Ένα θέμα που προκύπτει όλο και περισσότερο είναι ότι το 2012 θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε το, το πρώτο στάδιο του προγράμματος για also here, uh, του ενιαίου ουρανού. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τι θα πρέπει να κάνουμε για την πρόθεση αυτού του προγράμματος και για το πακέτο για, τη, για, το, το, για τους σιδηροδρόμους θα είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα του χρόνου για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες δράσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. So, if I can start... Λοιπόν, να ξεκινήσω με τους συντονιστές και μετά θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής για κάποια απάντηση. Τέσσερα λεπτά θα δοθούν στους συντονιστές και ίσως τρία λεπτά για τους υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Αλλά ως, αν όσο συμβεί συνήθως κάποια στιγμή σε μέσα συζήτηση κάποια άλλη στο λόγο, θα αλλάξει ο χρόνο που θα διατηθεί στον καθένα. Τέσσερα λεπτά καταρχάς στους συντονιστές. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σα παρουσιάσετε πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ένα συγκεκριμένα και δείτε την Λευκή Βίλη του 2010-2011. Το 2010 θα λάβουμε αυτό το έγγραφο εργασία. Θα το λάβουμε στο τέλος του χρόνου. Γιατί σίγουρα θα ήταν ενδιαφέρον. Εν τω μεταξύ διαβάζουμε διάφορα άρθρα τα οποία δημοσιεύονται στον τύπο που κάνουν διάφορε εικοσίε ό,τι αφορά το έγγραφο εργασία. Καλό θα ήταν λοιπόν να το έχουμε το συντομότερο δυνατό στα χέρια μα αυτό το έγγραφο εργασία. Η λευκή αυτή βίβλο, όπω ήδη συζητήθηκε και στα πλαίσια τη Επιτροπή αυτή και στην Ολομέλεια, εστιάζει σε κάποια θέματα τα οποία ήδη γνωρίζουμε και θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα κύρια θέματα. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, Ελπίζω όλες οι ευχές σας να ε, συγκεκριμενοποιηθούν. Η χρηματοδότηση των διαφορών διευρωπαϊκών δικτύων είναι σημαντική, αλλά πρέπει να συνεργαστούμε και με άλλες επιτροπές. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιου είδους συνεργασία. Το 2011 θα πρέπει να ληφθούν σαφείς αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά το πακέτο για τα αεροδρόμια, είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, το όλο πακέτο. Δεν θα επέκταθα από αυτού. Εν τω μεταξύ θέλω να θέξω άλλο ένα ζήτημα. Είναι σημαντικό να δούμε τι θα γίνει συγκεκριμένα και στο νομοθετικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, για το θέμα του ενιαίου ουρανού, δεν είναι αποδεκτό να συμβεί αυτό που συνέβη με το πρώτο πακέτο. για το ενιαίο δικό δικτύο. Προς το παρόν λοιπόν αφήνουμε όλη την ευθύνη, αλλά ξεκινάμε με την ε, υπόθεση ότι στη συνέχεια θα ενημερώνεται τακτικά το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τις ημερομηνίε, ε, τα ορόσημα που έχουν τεθεί σε ό,τι αφορά το πακέτο αυτό που αφορά και την κινητικότητα αλλά και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, εσωτερική αγορά, είναι η εσωτερική αγορά. Ίσως θα πρέπει να ανοίξουμε και για το άνοιγμα αυτής της αγοράς. Εν πάση περιπτώσει, δεν το έχουμε δει αντίστοιχα και, για τις, ε, και στις μεταφορές. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει κάποια σχετική νομοθετική πρόταση το 2012 ίσως. Ίσως κινούμαστε λίγο γρηγορότερα από εσά. Και το καμποτάζ είναι μεγάλο ενδιαφέροντος και θα συζητήσουμε τις ε, περαιτέρω εξελίξεις αυτού. Προφανώς όμως χρειαζόμαστε αξιόπιστες πληροφορίες σε σχέση με περιβαλλοντικές πτυχές. Και υπάρχει και το όλο θέμα των ε, ε, φορολογίας της, των τελών κυκλοφορίας ευρωβινιέτας και το θέμα επίσης των υπηρεσιών ταχυδρομείων που έχουν ζητηθεί και στο παρελθόν. Πάντα είμαστε σε τελική φάση. Πρέπει και αυτό να το δούμε. Και αν μιλάμε για ολοκλήρωση εταιρική αγορά, νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να δούμε τα επερχόμενα χρόνια και ο, ο ρόλος των διαφόρων ε, υπηρεσιών ανά την Ευρώπη. Χαίρομαι ότι αυτά που είδαμε στο παρελθόν και έχουμε σαφή ανάλυση για τις διάφορες υπηρεσίες και παρατηρητήρια στο πώς λειτουργούν, θα το εξετάσουμε πρωτού προχωρήσουμε στην θέσπιση και ε, στην εγκατάσταση νέων υπηρεσιών. Συμφωνούμε με την πρόταση σε ό,τι αφορά την υπηρεσία σιδηροδρόμων, γιατί θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εναρμόνιση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Αλκαντζόη, δύο λεπτά, για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε, σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Συμφωνούμε μαζί σας ότι το πρόγραμμα εργασίας ε, περιέχει μια σειρά πρωτοβουλειών, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει περισσότερα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να οδηγήσει φακέλους προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένες ε, επενδύσεις και κατευθύνσεις γραμμές σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά δίκτυα και ως Επίτροπος πρέπει να εφαρμόσετε η φυστάμενη νομοθεσία, υπάρχουν πτυχές επιτροπολογίας κλπ. κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να τύχουν ενιαίας διαχείρισης για να επιτύχετε τους στόχους σας. Και έτσι έρχομαι στη Λευκή Βίβλο. Θα πρέπει να αποτελέσει την βάση πολιτικής για τα επερχόμενα χρόνια. Είναι ένα σημαντικό έγγραφο στρατηγικής αλλά πραγματικά σας απευθύνω την πρόκληση να κάνετε κάτι πιο δυναμικό θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο και να αναφέρει χρηματοοικονομικά ή νομοθετικά μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τα επόμενα έτη. Διαφορετικά θα είναι μια καινή συζήτηση. Και έρχομαι σε κάποια σχετική κριτική. Αυτό που βρήκαμε εξαιρετικά σημαντικό στο κοινοβούλιο αυτό είναι ότι αναγγέλλεται αυτό το οποίο σκοπεύετε να πράξετε, όμως θα πρέπει ταυτόχρονα και να ε, πράξετε και να εφαρμόσετε αυτά που έχετε αναγγείλει. Και νομίζω ότι η Λευκή Βίβλος θα πρέπει να εμφανιστεί κάπου Ιανουάριο-Φεβρουάριο, γιατί ήδη είχε αναγγελθεί για τον Νοέμβριο. Και αυτό ισχύει και για αρκετά άλλα παιδεία. Επί σειρά ετών συζητάμε, για παράδειγμα, τα θέματα κατανάλωσης του, ε, προστασία συγγνώμη, του καταναλωτή. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πει ότι θα έπαιρνε κάποια νομοθετική πρωτοβουλία το 2010 για περίπτωση πτώχευση τραπεζών, παραδείγματι. Δεν έχουμε κάτι σχετικό από εσά. Είναι σημαντικό να τηρούνται οι ημερομηνίε που έχουν αναγγελθεί, που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Είπατε μια σειρά πραγμάτων που πρέπει να γίνει ολόκληρη εσωτερική αγορά. Συμφωνούμε ω ομάδα και το υποστηρίζουμε, αλλά και αυτό θα πρέπει να συμπορευθεί με κοινωνική πολιτική, καλή καταναλωτική προστασία και παροχή υπηρεσιών. Όλα αυτά έρχονται σε ένα πακέτο. Ο ενιαίος ε, ουρανός. Συμφωνώ μαζί σας. Υπήρξε πληθώρα φήμων που κυκλοφόρησαν ότι τα κράτη-μέλη ουσιαστικά χρονοτριβούν. Η νομοθεσία όμως έχει εφαρμοστεί. Υπάρχουν καταληκτήριες ημερομηνίες. Πρέπει να πούμε λοιπόν ό,τι είναι δυνατόν για να τηρήσουμε αυτές τις ημερομηνίες. Η μεταρρύθμιση των δρόμων είναι ένας άλλος σημαντικός φάκελος, όπου και πάλι επαναλαμβάνω ότι πρέπει να ανοίξουμε την αγορά, αλλά και πάλι για να έχουμε σωστή πολιτική σιδηροδρόμων. Και αυτό συμβαδίζει με την προσέγγιση των συνδυασμένων μέσων μεταφοράς και της κοινωνικού χρημα... Ε, μηχανισμού χρηματοοικονομικής ε, στήριξης. Ενδιαφέρονται λοιπόν διάφορα θέματα που έχουν τεθεί θα κοιτάξουμε να έχουν όλοι παρακολουθεί και ελπίζουμε να έχετε το σθένος, να επιτύχετε όλα αυτά που έχετε ανακοινώσει και ελπίζουμε να τύχετε και τις υποστήριξη των κρατών μελών. Γιατί πολύ συχνά τα κράτη-μέλη χρονοτριβούν πραγματικά σε ό,τι αφορά και ε, χρονοτριβούν και βάζουν φρένο. Ευχαριστώ που μας παρουσιάσατε το πρόγραμμα εργασίας για τη χρηματοδότηση των υποδομών. Ελπίζουμε όλοι ότι θα λειτουργήσει το σύστημα και θα βρούμε τα αναγκαία κεφάλαια. Αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο, πιστεύω. Και οι συζητήσεις σας με τους άλλους επιτρόπους ελπίζουμε ότι θα ευωδώσουν και θα οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Μιλήσατε για τα δικαιώματα των επιβατών και για αυτό το θέμα ελπίζω ότι θα τα εξασφαλίσουμε αυτά τα δικαιώματα πρόκειται, και ε, πρόκειται να γίνει αυτό στη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας για το άνοιγμα της υδροδρομικής αγοράς στην Ακρόαση. Είχατε πει ότι αυτό είναι σημαντικό για εσάς αλλά και για μας για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς για το σύνολο της Ευρώπης. Στείλετε μια ε, επιστολή σε ορισμένα κρατημέλη λέγοντάς ότι δεν είχαν κάνει τη δουλειά τους σε σχέση με το σιδηροδρομικό πακέτο. Έχουν επανέλθει στην τάξη. Ποιες ήταν οι συνέπειες αυτής της επιστολής. Δεν μιλήσατε για το e-ticketing. Είπατε ότι πρέπει να δίνονται καλύτερες πληροφορίες στους ε, επιβάτες για τη χρήση των σιδηροδρόμων. Αυτό το έχουμε τονίσει κατά επανάληψη μπορούμε να προβλέψουμε ηλεκτρονικά εισιτήρια για τα αεροπλάνα, αλλά όχι για τους σιδηροδρόμους. Μας είπατε ότι θα το κάνετε αυτό και θα θέλαμε πιο πολλές πληροφορίες. Και έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση ε, ε, τώρα. Τι δυνατότητες για το θείο και το άζωτο και τις εκπομπές τους στη Βελτική ειδικότερα. Πρέπει να μην υπάρξει στρέβλωση του ανταγωνισμού πρέπει να γίνουν σεβαστοί ορισμένοι κανόνες για τα επόμενα χρόνια. Πρέπει, καλό είναι να έχουμε φιλόδοξους στόχους, αλλά η έκθεσή μου για τη θαλάσσια πολιτική δεν το είχε λάβει τότε υπόψη, αλλά τώρα τι γίνεται με τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε θα υπάρχει παντού προστασία του περιβάλλοντος χωρίς υπερβολές με αποτέλεσμα να, επηρεαστούν δυσμενώς οι σιδηροδρομικές μεταφορές. Για την Οροβινιέτ. Λυπάμαι και θα συμφωνήσετε φαντάζομαι μαζί μου ότι για την Οροβινιέτ θα μπορούσαμε να είχαμε εξασφαλίσουμε ε, μια χρηματοδότηση από τις υποδομές με τα έσοδα της εσωτερικοποίησης των εξωτερικών δαπανών, αλλά δεν λειτουργεί σε αυτό το σύστημα. Έχω ακόμα μερικά δευτερόλεπτα στη διάθεσή μου για τα αεροδρόμια. Οι εμπορευματικέ μεταφορές, αεροπορικές μεταφορέ, η, αεροπορική, μεταφορά, αεροπορική μεταφορά εμπορευμάτων, γι' αυτό μα είπατε ότι θα δείτε ποιε βελτιώσει πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν κανονισμοί, του οποίου συζητήσαμε σήμερα το πρωί, σε τι μέτρο ε, γίνονται σεβαστοί και εφαρμόζονται. Η Επιτροπή μας είπε ότι από τον Απρίλιο 2011 τα υγρά θα ελέγχονται δεν ήταν αυτό που είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο. Εμείς θέλαμε να υπάρχουν ειδικέ σακούλες για τις αγορές που γίνονται στα καταστήματα των ειδών. Μια ενδιάμεση λύση προτείνουμε να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούνται σαρωτές, ότι αρκούν οι σακούλες. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω πότε θα εμφανιστεί αυτή η, λευκο, η λευκή βίβλος. Στο τέλος αυτού του έτους, στο προσεχές, θα ήθελα να το ξέρω. Αποφασιστική σημασίας βεβαίως είναι και το κόστος. Θέλουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον, αλλά θέλουμε να ξέρουμε πώς έχει η οδική ε, υποδομή και ποιο είναι το ενεχόμενο Είπαμε ότι ένα 40% θα δοθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο και 60% στο οδικό. Θα αλλάξει αυτή η ποσοστία αναλογία ή όχι. Ποια θα είναι τα ποσοστά ή τα κονδύλια όταν μιλάμε για τα μεγάλα σιδηροδρομικά προγράμματα. Έχουμε τα αναγκαία κονδύλια ή σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τα μικρότερης εμβέλειας σχέδια για την ε, αναμόρφωση των σιδηροδρόμων. Τι θα γίνει ως προς τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρόμων. Δεν μπορούμε να έχουμε διεθνή εισιτήρια εύκολα. Τι θα κάνετε σε σχέση με πέρσι, διότι πέρσι μιλήσαμε για ένα σιδηροδρομικό πακέτο το οποίο ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί από όλα τα κράτη-μέλη και θα ήθελα να ε, ρωτήσω γιατί δεν έχει εφαρμοστεί αυτό το πλαίσιο ως προς την μείωση των ε, ανισορροπιών ή των ανισοτήτων ε, γενικότερα. Δεν θα μπορούσατε να κάνετε κάτι και στον τομέα των ε, σιδηροδρόμων, δηλαδή οι επιβάτες να μπορούν να λαμβάνουν αντισταθμίσεις, όπως ισχύει στην αεροπλοεία. Όταν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, δεν θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ όλων των μέσων μεταφοράς. Ως προς την ε, τεχνολογία στους ε, σιδηροδρόμους, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές επιχειρήσεις δεν μπορούν να πουλήσουν τους νέους σύρμους που διαθέτουν, διότι πολλές φορές οι οικονομικοί φορείς ε, προτιμούν τους παλαιότερους σύρμους από τους νέους. Τι προβλέπετε σε αυτή την περίπτωση. Πώς μπορείτε να υποστηρίξετε τις επιχειρήσεις οι οποίες προβάλλουν νέα προϊόντα στην αγορά. Βεβαίως μιλάμε για την προστασία του περιβάλλοντος, μιλάτε για το θαλάσσιο πακέτο, όμως γνωρίζουμε ότι στα μεγάλα πλοία δεν προβλέπονται ειδικά φίλτρα προστασίας. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα. Τι θα γίνει ως προς το θαλάσσιο πακέτο σε σχέση με τη χρήση κινητήρων. Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον Επίτροπο για την παρουσίαση. η Λευκή Βίβλος θα δημοσιευθεί λίγο αργότερα από ό,τι είχε ανακοινωθεί, αλλά κατά μένα δεν είναι και το τραγικό. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που ανέφερε ο Επίτροπος, ότι δηλαδή θα είναι ένα στρατηγικό έγγραφο που θα οργανώνει τις ε, μεταφορές και την ενέργεια. Είναι σωστή η προσέγγιση κατά την μου, γιατί θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε και να καλύψουμε αυτή την ανάγκη χρηματοδότηση στην επόμενη περίοδο. Επί των θεμάτων που ανέφερε ο Επίτροπος, θα ήθελα να αφαιρθώ στα δικαιώματα των επιβατών. Ήδη έχουν αναπτύξει άλλοι το θέμα αυτό, αλλά καλό θα ήταν να ε, πάρουμε κάποια μαθήματα από την κρίση με την ηφαιστειακή τέφρα για να βελτιώσουμε τη σχετική νομοθεσία προστασίας των επιβατών. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική έκδοση ε, εισιτηρίων, το e-ticketing είναι βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι των δικαιωμάτων των επιβατών. Χωρί τη σχετική νομοθεσία θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στο project αυτό. Μπορούμε να πάρουμε λοιπόν το παράδειγμα από την αεροπλοεία σε ό,τι αφορά το e-ticketing. Σε ό,τι αφορά τις ε, μεταφορές φορτίων, ίσως θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε την πρόοδο που υπάρχει στο πεδίο των χρονικών περιόδων, των slots που υπάρχουν. Εξακολουθεί να υπάρχει ο κανόνας, χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο slot, το χρησιμοποιήσει, το χάνεις. Ποια είναι η ιδέα σε ό,τι αφορά επίσης τη σχετική οδηγία για τον επίγειο χειρισμό των αποσκευών και για το καμποτάζ. Χθε είχαμε μια συζήτηση όταν συζητήσαμε για το θέμα του ανταγωνισμού. Θέλω να ακούσω την άποψή σας των θεμάτων, των εμποδίων που υπάρχουν για το καμποτάζ, γιατί γίνονται διάφορες αντιρρήσεις από τα κράτη-μέλη. Φορείς ε, από διάφορα κράτη-μέλη ε, εφαρμόζουν στρατηγικές dumping, ακόμα και στο κοινωνικό επίπεδο, για να αντιταχθούν στο καμποτάζ. Ποια είναι η σχετική σας θέση. Προσπαθούμε να καθιδρύσουμε αρχές ισότιμης ε, διαχείρισης και αντιμετώπισης στην εσωτερική αγορά. Εάν λάβουμε όμως υπόψη τις διαφορές μισθοδοσίας, κάποιες χώρες ε, είναι, όταν πληρώνουν πολύ χαμηλότερα και από τον ελάχιστο δυνατό μισθό, δεν θα μπορούν πουδενή να ανταγωνιστούν σε ισότιμη μεταχείριση των τρανς. Και δεν μιλάω για την εφαρμογή των κανόνων στις ε, βαριές μεταφορές, όπως για παράδειγμα την παραβίαση των ε, ορών οδήγησης κλπ. Πάλι θα υπάρχει αντίστοιχο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υποβάλω τρεις ερωτήσεις μόνο. Πρώτον, σε όλες τις ε, συμφωνίες προσχώρησης αναφέρεται το καμποτάζ. Κύριε Επίτροπε, τι θα κάνουμε με το καμποτάζ. Αυτή είναι μια ερώτηση που μας ενδιαφέρει, που ενδιαφέρει όλες τις χώρες που προσχώρησαν πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για παραβίαση των θεμελιωδών ελευθεριών και πρέπει να εξασφαλίσουμε εν, ίσους, ίσους κανόνες για όλους σε αυτό το τομέα. Και κάτι που δεν αναφέρθηκε εδώ, για τα άτομα με αναπηρίες υπάρχουν σαφείς εικόνες, σαφή εικονίδια που χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη. Αυτά τα εικονίδια, ωστόσο, δεν είναι αναρμονισμένα σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι που θα έπρεπε να γίνει. Μπορείτε να κάνετε κάτι, είναι ένας τομέας που αγνοείται για πάρα πολύ διάστημα. Άτομα με αναπηρίες, όταν χρησιμοποιήσουν μια κάρτα που έχει εκδοθεί στην Τσεχία, θα χρειαστεί να πληρώσει ε, πρόστιμο αν παρκάρει κάπου το αυτοκίνητό του στην ε, Πολωνία, επειδή δεν χρησιμοποιεί την κατάλληλη κάρτα, παρόλο που τα εικονίδια είναι παντού, θα έπρεπε κανονικά να είναι παντού τα ίδια. Χρειάζεται λοιπόν ένα αρμόνι στον κανόνα. Λοιπόν, θα απαντήσετε στην πρώτη ομάδα των ερωτήσεων από τους συντονιστές και υπάρχει και ένας μακρύς κατάλογος ομιλητών για το δεύτερο γύρο. γύρο. Ωραία. Θα Προσπάθησα να ομαδοποιήσω αυτά τα θέματα. Το θέμα της Λευκής Βίβλου είναι ένα από τα θέματα στα οποία αναφέρθηκαν οι περισσότεροι ομιλητές. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι βρίσκεται στο τραπέζι μου, στο γραφείο μου αυτή τη στιγμή. Και μια τέτοια λευκή βίβλος, σκοπός μας είναι να περάσει από όλες τις διαδικασίες ε, τις ενδοϊπηρεσιακές, όλες τις συζητήσεις κλπ. Και αυτό θα πετύσει χρόνο. Αλλά στη διάρκεια αυτού του έτους και πριν έχετε το κείμενο στα χέρια σας, αυτό είναι που θα προσπαθήσω να κάνω να ετοιμάσω ένα concept paper δηλαδή που θα είναι σύντομο, 10-15 σελίδες θα έχει και αυτό θα, θα είναι ο πυρήνας, ο πυρήνας της δράσης μας. Πρέπει να πω ότι στον τομέα των μεταφορών γίνανε πολλά καλά πράγματα φέτος. Δεν τα πήγαμε και τόσο άσχημα. Το θέμα της Ροβινιέτ πέρασε πέρασε από το Συμβούλιο με μια πάρα πολύ μικρή αναστέλουσα μειοψηφία και στις ακροάσεις είχα ρωτηθεί ποιες είναι οι προοπτικές. Ε, έγινε το πρώτο βήμα και θα ε, προχωρήσουμε με τη χρηματοδότηση και όλα τα άλλα. Το Δεκέμβριο θα υπάρχει πλέον αυτή η εφαρμογή, διασυνοριακή εφαρμογή ε, προστήμων και ποινών για παραβάσεις της, του, του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Θα καταβάλω πάρα πολλές προσπάθειες να γίνουν όλα αυτά, διότι είναι κάτι που το περιμένει η κοινότητα των μεταφορέων και οι πολίτες. Οι δράσεις που προβλέπονται για τα επόμενα χρόνια αναφερθήκατε στο θέμα του ενιαίου ουρανού και ποιο είναι το πρόβλημα ρωτήσατε. Το πρόβλημα είναι ότι τα κράτη-μέλη αποφάσισαν ότι υπάρχουν δύο εναλλακτικέ λύσεις για να προχωρήσουμε, ε, να προωθήσουμε αυτό το πρόγραμμα του ενιαίου ουρανού. Από πάνω προς τα κάτω, να ετοιμάσουμε δηλαδή ένα νέο πρόγραμμα. Αυτό ομόφωνα απορρίφθηκε από τα κράτη-μέλη και μια δεύτερη πρόταση έγινε δεκτή, μια πρόταση που ξεκινά από τη βάση και, πηγαίνει προς τα πάνω, δηλαδή τα κράτη-μέλη δέχθηκαν να, γίνει, να υπάρξει μια δοκιμαστική περίοδος προτού καθιερωθεί ο σύστημα. Την περασμένη εβδομάδα περίπου έγινε μια συνάντηση ε, εκπροσώπων των κρατών μελών οι οποίοι αρνήθηκαν, απέρριψαν κάποιες ε, ε, πλευρές αυτής ε, της πρότασης. Αυτό που περιμένει από εμά η αεροπορία είναι ότι αυτό το πρόγραμμα του ενιαίου ουρανού θα προχωρήσει, θα υλοποιηθεί. Στο Συμβούλιο Μεταφορών αρχές Δεκεμβρίου ελπίζω να συζητηθεί αυτό το θέμα και όσον αφορά και αν η προσέγγιση με βάση τις επιδόσεις δεν προχωρήσει, θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι άλλο για του χρόνου. Για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Η αναμόρφωση της πρώτης δέσμης μέτρων ήταν περιορισμένη. Υπάρχει προθυμία και σε επίπεδο επιχειρήσεων και είχα πολλές επαφές να προχωρήσουμε με ένα αποτελεσματικό πακέτο που θα, κάνει, που θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα των σιδηροδρόμων ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν τις οδικές μεταφορές. Διότι με τη σημερινή κατάσταση, τον κατακαιρματισμό που υπάρχει τώρα, αν συνεχιστεί δεν θα γίνει τίποτε. Ελπίζω λοιπόν θα μπορέσουμε του χρόνου να παρουσιάσουμε ε, προτάσεις ε, για την πιστοποίηση του τροχαίου υλικού και πρέπει να δώσουμε στην αρμόδια υπηρεσία ευρύτερες αρμοδιότητες για να ασχοληθεί με αυτό το θέμα της δυνατότητας πρόσβασης ε, στις υποδομές των σιδηροδρόμων, στις ε, σιδηροτροχές. Με βάση αυτό το πρόγραμμα πιστοποίησης. Αυτές είναι οι σημαντικές δράσεις που σκοπεύουμε να αναλάβουμε έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες κατά 22 κρατών μελών επειδή δεν εφαρμόζουν τον κανονισμό, τον κανονισμό για τους σιδηροδρόμους. Το θέμα τώρα των ηλεκτρονικών εισιτηρίων είναι κάτι το ενδιαφέρον για τους σιδηροδρόμους. Υπάρχει το θέμα των τεχνικών προδιαγραφών για τη διαλειτουργικότητα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τηλεματικών λύσεων για την εξυπηρέτηση των επιβατών ε, την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των επιβατών. Είναι περίπλοκη η ονομασία αυτή. Αυτό που έχει σημασία είναι να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα ε, για τις σιδηροδρομικές μεταφορές ανάμεσα στα διάφορα κράτη. Πρέπει να προταθούν συγκεκριμένα πρότυπα και αυτό σκοπεύουμε να προωθήσουμε. Τώρα το θέμα του IMO, του Παγκόσμιου Οργανισμού Ναυτιλίας. Όταν θα θεσπιστεί η νομοθεσία δεν θα υπάρχει δυνατότητα υπαναχώρησης στη Νότια Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Τι θα γίνει. Είναι ένα θέμα σημαντικό για το οποίο πρέπει να προτείνουμε κάποιους δίκαιους κανόνες. Τα υγρά. 2013 πρέπει να ελέγχονται, να σαρώνονται. Υπάρχει τώρα η σχετική τεχνολογία. Όταν αναφέρθηκε πρώτη φορά αυτό το θέμα, ελέγχθη ότι κάτι πρέπει να γίνει για να μην χρειάζεται οι άνθρωποι να κουβαλάνε ε, τα υγρά που μεταφέρουν, αλλά να υπάρχει δυνατότητα σάρωσης όταν βρίσκονται μέσα στις αποσκευές τους. Αναζητούμε λοιπόν τις καλύτερες δυνατές λύσεις από για το 2013 και πέρα. το νέο πρόγραμμα για, τις διευρωπαϊκές, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ε, στον τομέα των μεταφορών ε, προωθείται. Δεν ξέρω πού ακριβώς έχουμε φτάσει ε, για το θέμα του φιλτραρίσματος του νερού. Για τα σλότς και τις χρονοθυρίδες πρέπει να εξασφαλίσουμε έναν πιο ευέλικτο χειρισμό τους αλλά δεν μπορώ να σας δώσω σήμερα λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Και ένα σημαντικό ενδιαφέρον θέμα έθεσαν δύο ομιλητές για το καμποτάζ. Η χώρα μου ε, ε, έχει επιβάλει τους ίδιους περιορισμούς για το καμποτάζ. Δεν είναι λοιπόν κάτι που αφορά μόνο τα νέα κράτη-μέλη, αλλά και τα παλιά θέλουμε να καταργήσουμε αυτούς τους κανόνες, γιατί αυτοί οι κανόνες για το καμποτάζ είναι κάπως απαρχαιωμένοι. Ήδη σήμερα, τρεις φορές την εβδομάδα, μπορείς να προσφέρεις υπηρεσίες. Και αυτό καθιερώθηκε για να καταπολεμηθεί ο φοβερός ε, φόβος, ο τρομερός φόβος για τον ανταγωνισμό αλλά που δεν επιβεβαιώθηκε, πρέπει λοιπόν να καταργηθούν αυτοί οι κανόνες. Και θα εκπνεύσουν, θα εκπνεύσουν εν πάση περιπτώσει. Δεν θυμάμαι πότε, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε ε, να έχουμε πια περιορισμό για το καμποτά στην Ευρώπη. Είναι μια απαρχαιωμένη ιδέα αυτή και εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που ήδη έχει αρχίσει να γίνεται. Νομίζω ότι κάλυψε τα περισσότερα από τα θέματα που ε, ε, προέκυψαν μέχρι στιγμής. Ευχαριστούμε δεύτερη σειρά μιλητών. Παρακαλώ πολύ περισσότερο στα δύο λεπτά. Οι πάντες μπορούν να παρέμβουν. Ο κύριος Κάντσον. Ευχαριστώ και από πλευρά μου, κύριε Επίτροπε. Προφανώς είναι εξαιρετικά χρήσιμες στιγμές για να κάνουμε και ένα σχετικό προγραμματισμό στο εταιρικό τη Επιτροπή μα. Ομολογώ όμω ότι είμαι εξαιρετικά ανήσυχο, κύριε Επίτροπε. Γιατί η χρόνη πολιτική, δυστυχώ αυτή τη ιδιαίτερη συγκυρία, είναι εξαιρετικά διαφορετική από του χρόνου που περίμενε ο κόσμο στην πράξη. Δεν ξέρω, όλοι κινούμεθα, αν θέλετε, στο πεδίο μα και διαπιστώνουμε μια, βλέποντα μακροσκοπικά την κατάσταση σε επίπεδο ανεργία. είναι ένα μείζον κοινωνικό θέμα ένα θέμα που πιέζει και έχουμε το καθήκον να προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε για αντιμετώπιση του. Σας ζητώ λοιπόν και σας κάνω έκκληση ώστε οι χρόνοι, το όλο timing να βραχυνσούν. Δεν είναι δυνατόν να βρισκόμαστε ακόμα στον απαρίθμηση του τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει ανυπερθέτως να υλοποιήσουμε το συντομότερο δυνατόν, το πιο σύντομο χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων που αναφέρεται. Ένα άλλο θέμα. Μιλάμε κατά κόρον περί προγραμματισμού. Δεν άκουσα καθόλου και δεν βλέπω τίποτα περί της ουσίας που θα πρέπει να είναι σε συσχετισμό με τον προγραμματισμό για να γίνουν επιχειρησιακά και λειτουργικά κάποια σχέδια. Η δική σας αναφορά και η λειτουργία σας είναι πάρα πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά τις υποδομές, γιατί σήμερα προσπαθούμε να εκφύγουμε από την κρίση αυτή πέρα από τα κοινωνικά κριτήρια που χορηγούνται, η υλοποίηση των έργων υποδομής είναι μια υλοποίηση μεγάλων προγραμμάτων ενέργειας, τουρισμού κλπ. Έχετε πολύ σημαντικό ρόλο λοιπόν κύριε Επίτροπε να διαδραματίσετε. Σας ζητώ λοιπόν αν από άποψη υλοποίηση υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο που θα μπορούσατε να μας πείτε και σε ό,τι αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές και τον προσανατολισμό, και τα κυρίαρχα στοιχεία που υπάρχουν για να μπορέσουμε να κάνετε αυτό που σας ζητώ, θα σας παρακαλούσα να προσπαθήσετε να αρχίσετε να εργάζετε άμεσα, ώστε να τον πιο γρήγορα λοιπόν και τη υλοποίηση. Αυτό έχω να ζητήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λάικφριντ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ένα ερώτημα έχω να υποβάλω και αφορά σε κάτι που άκουσα, γιατί υπάρχουν κάτι πολύ δυσάρεστες φήμες που κυκλοφορούν είναι το θέμα Gigaline. Πέρσι, την τελευταία περίοδο, ε, λύθη μια πολύ καλή απόφαση του πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των μεγάλων υπεροκινιανίων που μπορούν να αποφασίσει κάθε χώρα να τα θέλει ή όχι. Τώρα ακούω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι φαίνεται να είναι υπέρ απαραίτητων αλλαγών. όντω ισχύει κάτι τέτοιο? Εάν ναι, και ελπίζω όχι, οφείλω να ομολογήσω, τι σκοπεύετε να κάνετε σε σχέση με τα πολύ μεγάλα υπεροκειάνια. Ευχαριστώ, κυρία Σάβησα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα μιλήσαμε για την ασφάλεια της αεροπλοείας και ιδιαίτερα Μιλήσαμε για τους αρωτές ε, σώματος. Νομίζω ότι η Επιτροπή Μεταφορών άρχισε να ασχολείται με θέματα ε, τρομοκρατίας, το οποίο είναι σημαντικό ε, βεβαίως, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να αφορά αυτή την Επιτροπή πάντα. Το θέμα είναι περισσότερο φιλοσοφικό, γιατί μιλάμε για ανθρώπους. Βεβαίως και οι τρομοκράτες είναι άνθρωποι και αν και θεωρούμε ότι δεν είναι και τόσο εφή ε, άτομα, όσο αυτοί που δημιουργούν τους αρωτές θα πρέπει να μας απασχολήσει κατά πόσο υπάρχει κάποια συνεννόηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πόσο μακριά μπορούμε να κινηθούμε σε αυτό τον ε, τομέα ασφαλείας για τα αεροδρόμια, διότι είναι μία ιστορία χωρίς τέλος. Ένας δημιουργεί μια μηχανή, ο άλλος την καταρρύπτει. Μετά ξαναδημιουργεί, ξανακαταρρύπτει. Πού υπάρχει το όριο, υπάρχει κάποιο όριο. Λίχτεμπεργκερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Καταρχήν, ένα ερώτημα ασχολούμαι, βρίσκομαι και στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και μιλάμε για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα και αποτυχία ως προς τον τομέα των μεταφορών. Και ένα από τα προβλήματα είναι ο χρόνος διακοπής εργασίας για τους οδηγούς. Ορισμένα κράτη-μέλη δεν έχουν εισαγάγει ελέγχους ο προκάτοχός σας είχε πει ότι θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Θα αναλυφθεί κάποια συγκεκριμένη δράση. Νομίζω ότι υπάρχουν κανόνες ανταγωνισμού βεβαίως, αλλά η Επιτροπή θα πρέπει να επιβάλλει ένα κοινό πλαίσιο. Όταν μιλάμε για κοινωνικά δικαιώματα δεν συμβαίνει τίποτα τόσο γρήγορα. Δηλαδή, για τους κανόνες ανταγωνισμού ε, η δράση είναι άμεση, αλλά ως προς το κοινωνικό όχι και τόσο, διότι μιλάμε για επιχειρήσεις κυρίως. Υπάρχουν έλεγχοι από μερικές επιχειρήσεις και από άλλες όχι. Θα ήθελα λοιπόν κάτι να κάνετε κύριε Επίτροπε και σε αυτό το τομέα έτσι ώστε να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος για πράγματα που έχουμε προαποφασίσει και που έχουμε εισαγάγει μαζί με το Συμβούλιο. Ε, πρόκειται για μία ε, πόδινη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Ε, αν τα κράτη-μέλη δεν κάνουν αυτά που πρέπει, τότε θα υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός στις οδικές μεταφορές και θα, πλήττουμε, θα πλήττονται οι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις. Και το μιλάμε και για την ασφάλεια. Ε, την οδική ασφάλεια. Κύριε Φώστερ, για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τα σχόλιά σας και τις πληροφορίες. Ευπρόσδεκτες βεβαίως οι, οι προτάσεις για τους σιδηροδρόμους, ιδιαίτερα για το ε, σύστημα έκδοσης εισιτηρίων, διότι βλέπουμε ότι πολλοί που θέλουν να ε, ταξιδέψουν Ευρώπη δεν μπορούν να εκδώσουν ένα εισιτήριο όταν θέλουν να μεταβούν από το βορρά στο νότο της Ευρώπης. Ελπίζω να το προωθήσετε αυτό. Σε σχέση με τα σχόλιά σας για το πακέτο αεροδρομίων και θέματα χρόνων, χρονισμού, όταν είδα την αναθεώρηση του κανονισμού των χρονοθυρίδων, ε, το θέμα ήταν ιδιαίτερα λεπτό Ελπίζω να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικός και για την αναθεώρηση του κανονισμού ε, ε, ε, ηχορύπανσης στην αεροπλοεία, δηλαδή η χορύπανση από τους κινητήρες θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Θα πρέπει να δούμε βεβαίως και το κόστος, που, το, το εμπλεκόμενο κόστος για τις βιομηχανίες. είδα ένα αρχικό σχέδιο του, της Λευκής Βίβλου, είναι λυπηρό ότι μέσα στις 200 σελίδες υπάρχει μία σελίδα μόνο για τον τομέα της αεροπλοείας. Και τότε δεν γινόταν μία στο SSR. Α, μιλήσαμε για, τους, για τον ενιαίο ουρανό 10 χρόνια πριν. Μιλάμε για το περιβάλλον, το κόστος, την αεροπλοεία, τον εναέριο χώρο γενικότερα. Και δεν είμαι καθόλου ευτυχής γιατί λέτε ότι αυτό θα συζητηθεί του χρόνου. Η βιομηχανία, ξέρετε ε, ότι, στο, ότι το Σέζαρ και δεν μιλάμε ε, παρά για το γεγονός ότι μόνο Δύο προγράμματα υπάρχουν. Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη όθηση από τα κράτη-μέλη. Το πρόγραμμα Caesar θα πρέπει να λειτουργήσει έμπρακτα. Θα ήθελα λοιπόν να ακολουθήσετε πιο σκληρή γραμμή ε, έναντι των κρατών μελών έναντι, ως προς το πρόγραμμα ΣΥΖΑΡ. Ε, Ο κύριο Κουμουτσάκος για δύο λεπτά. Κύριε Πέτροπε, ευχαριστώ για την ε, ενημέρωση που μα κάνατε σήμερα. Πηγαίνω κατευθείαν στο ερώτημά μου. Άκουσα με μεγάλη προσοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αναφορά σα στην κοινωνική ατζέντα για τους ε, ναυτικού. Και είναι δίκαιο για αυτού του ανθρώπου που δουλεύουν 24 ώρες 24 ώρο να προβλεφθούν και να ενταχθούν στην κοινωνική ατζέντα. Όμως κύριε Επιτρόπε πρέπει να σας ομολογήσω ότι δέχομαι με ορισμένα ανισχυτικά αντιφατικά μηνύματα από την πλευρά ε, της Επιτροπής. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πλευρά της Επιτροπής που ε, υποστηρίζει ορθώς να ενταχθούν οι ναυτικοί στην ε, κοινωνική ατζέντα, ειδικά όσον αφορά τη σύνταξή τους, ενώ άλλες πλευρές της Επιτροπής, άλλη διεύθυνση της Επιτροπής, η οποία μάλιστα προετοιμάζει μια σειρά οδηγιών ε, οριζόντιας ε, λογικής, ε, σκοπεύει ή, εν πάση περιπτώσει, επιθυμεί ή βλέπει ότι οι ναυτικοί πρέπει να ενταχθούν σε αυτές τις οδηγίες ε, σαν να μην υπάρχει καμία διαφοροποίηση για τους ναυτικούς από άλλους εργαζομένους και είναι ένα αντιφατικό μήνυμα που με προβληματίζει πρέπει να σας πω. Όσον αφορά για τα ζητήματα της ναυτιλίας, ε, είναι γνωστό κύριε Επίτροπε ότι πρέπει να διατηρήσουμε ειδικά στις σημερινές πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Πόσο μάλλον όταν υπάρχουν αναδυόμενες νέες δυνάμεις που έχουν κάνει τον διεθνή ανταγωνισμό ακόμα πιο σκληρό από ό,τι ήταν στο παρελθόν και μερικές φορές αθέμητο. Ε, επομένως και με δεδομένο ότι η ναυτιλία είναι, παραμένει ο πιο φιλικό τρόπο μεταφορά για το περιβάλλον, θέλω να σα ρωτήσω, γιατί ακούω ορισμένε απόψει για συμπερίληψη τη ναυτιλία στο σύστημα ETS. Πιστεύω ότι είναι μια εσφαλμένη θέση, κάνει κακό στην ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή ναυτιλία σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την ευρωπαϊκή οικονομία. Τέλο, όσον αφορά την τα κάψιμα με την περιεκτικότητα θείου, νομίζω ότι όλοι παραδέχονται ότι το όριο του 0,1 είναι απολύτω μη ρεαλιστικό. Αυτά τα καύσιμα είναι πανάκριβα και είναι περιορισμένα, εξαιρετικά περιορισμένα για να καλύψουν τις, ε, τις ανάγκες που υπάρχουν. Δεν επαρκούν με λίγα λόγια. Μάλιστα, κράτη τα οποία συμμετέχαν στη Συμφωνία της Βαλτικής έχουν τώρα δεύτερες σκέψεις και ορισμένοι έχουν ήδη μετανιώσει που συμμετέχουν σε αυτό. Θα ήθελα την άποψή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much, Mr. Λιβεράτσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Είμαι πολύ θετικά διακείμενος απέναντι στην παρουσίασή σας, αλλά θέλω να σε επισημάνω και το ακόλουθο ζήτημα. Το πρώτο είναι οι οικονομικές ε, συνθήκες των ε, Ευρωπαϊκών ε, Μεταφορών. Το δεύτερο είναι οι οικονομικές συνθήκες των εταιριών εφοδιαστικής και μεταφορικές. Νομίζω ότι θα άξιζε να αφιερώσουμε τη συνάντησή μας εδώ για να μιλήσουμε τα θέματα αυτά. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σε ό,τι αφορά την οικονομία. Ε, τις ε, συνολικές πτυχές, ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά, αεροπλοεία και ναυσιπλοεία. Και επίσης το σύνολο των μεταφορών και μεταφορικών εταιριών. Ίσως θα έπρεπε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες εργασίας και συνθήκες ε, πληρωμής των εργαζόμενων στον τομέα αυτό. Μιλάμε για τα δικαιώματα των επιβατών, αλλά θα έπρεπε να εξετάσουμε και τα εργατικά, τα δικαιώματα των εργαζομένων στο πεδίο, στον τομέα αυτό. Οι ναυτιλιακές μεταφορές, οι ζεδρομικές μεταφορές επίσης πρέπει να εξεταστούν και θα πρέπει να δούμε επίσης τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις από την εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους. Ίσως θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να δούμε το μέλλον του όλου ζητήματος. Και δύο ακόμα στοιχεία. Το ένα, η ενοποίηση των κανόνων χρήσης των δημόσιων μέσων μεταφοράς στην Ευρώπη. Εδώ βλέπουμε τις διαφορές σε ό,τι αφορά την υποδομή και το καθεξής. Και ένα άλλο θέμα, εάν θέλουμε να αποτιμήσουμε την εφαρμογή του πρώτου πακέτου για τις μετα... για τους αεροδρόμους, είναι ότι από τις 25 χώρες, στις 23 έχουμε μεγάλες παραλήψεις και παρεκκλήσεις. Μήπως πρέπει να θεωρήσουμε τους κανονισμούς, γιατί ίσως να υπάρχει υπερβολικό πλέγμα κανονισμός μεταφορές. Ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε καλύτερα την εφαρμογή των κανονισμών που έχουμε θεσπίσει. Ευχαριστούμε, κύριε Σασάλ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας συγχαίρω για το πολύ φιλόδοξο αυτό σχέδιο και χαίρομαι που τόσα πολλά θα αντιμετωπίσει και θα εξετάσει η Επιτροπή τόσο γρήγορα. Και είναι πολύ καλό που θέλετε να ασχοληθείτε με τα δικαιώματα των επιβατών σε ό,τι αφορά άλλον τρόπο μεταφορών, αλλά θα πρέπει να θυμηθούμε επίση ότι υπάρχουν και κάποιοι επιβάτε που ήδη χαίρουν των δικαιωμάτων του. Η εφαρμογή όμω των δικαιωμάτων είναι πρόβλημα. Και εδώ εννοώ, του υπονοώ τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα που κινούνται αεροπορικά και, δι, και επίσης τα άτομα που κινούνται με μικρά παιδιά. Οφείλω να αναφέρω εδώ ότι η εφαρμογή, η χρήση του κανονισμού 1107 πραγματικά αφήνει πάρα πολλά ανοιχτά θέματα. Και ένα άλλο θέμα είναι η υποτιμολόγηση κάποιων αεροπορικών εταιριών, οι οποίες κοστολογούν επιπροσθέτως εάν χρησιμοποιήσει την πιστοτική σου κάρτα για την πληρωμή του στηρίου σου. Ευχαριστούμε. Ε, κυρία Σέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με συγχωρείτε, έπρεπε να βγω διότι όπως ξέρετε έχουμε μεγάλα προβλήματα στην Επιτροπή Αναφορών και έπρεπε να βγω για μία συγκεκριμένη αναφορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κάλας για την παρουσίαση αυτή. Θα ήθελα απλώς να αναφερθώ στην παρουσίαση του κειμένου της Επιτροπής ως προς το πρόγραμμα Μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη και για smart growth γενικότερα και στον τομέα των μεταφορών. Μιλάμε για την ενέργεια, θέματα μεταφορών και ε, θέματα γεωργίας. Και βλέπω ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις. Δεν ξέρω κατά πόσο στα πλαίσια της ενέργειας μπορούμε να μιλήσουμε για απασχολησιμότητα και καινοτομία. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια κρυπτογραφική γλώσσα ως προς τις μεταφορές. Δηλαδή δεν προσεγγίζουμε τον πολίτη χρησιμοποιώντας αυτή την ιδιόγλωσσα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Επίτροπε, ποιες πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει στον δημοσιονομικό τομέα και τι θα μας προτείνετε για το 2011, πόσες πρωτοβουλίες νομοθετικού περιεχομένου λοιπόν για το 2011 και τι ποιο προϋπολογισμό προβλέπετε για τα δίκτυα. Για να δούμε και τις δημοσιονομικές πρόπτικες από το 2013 και μετά. Διότι όπως ε, ξέρετε ε, υπάρχουν όρια στο σχέδιο Γαλιλαίο και θα θέλαμε να ξέρουμε τι σκέφτεστε έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας υποστηρίξουμε. Πότε θα μας μιλήσετε για τα δίκτυα. Ως προς τα δικαιώματα των επιβατών χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συνοχή και μία πρόταση της Επιτροπής που να έχει αυτή την ε, ομοιογενή σφαιρική προσέγγιση για όλα τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να μην υπάρχουν διαφορές ως προς τις μεταφορές. Ως προς τις οδικές μεταφορές θα ήθελα να σας πω πού υπάρχουν θέματα αστικής κινητικότητας, πώς τοποθετούμε την ατζέντα μεταφορών και τι θα κάνετε ως προς την επιμελητιακή ε, βοήθεια, την τεχνικοηλική βοήθεια για τις διατροπικές μεταφορές. Τέλος, Επίτροπε, να πω κι εγώ δύο-τρία πράγματα για να τα λάβετε υπόψη προτού απαντήσετε στις ε, πολλές παρεμβάσεις του δευτέρου γύρου. Για τα τεντή πρέπει να δούμε ε, τον, τον καθορισμό προτεραιοτήτων αυτών των έργων. Με έμφαση έχουμε πει ότι θα θέλαμε οι διασυνοριακές συνδέσεις και τα σχετικά προβλήματα να επιληθούν καθώς και όλα τα άλλα σημαντικά προβλήματα που ε, προκύπτουν στον τομέα των μεταφορών. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία για το e-ticketing, για τα ηλεκτρονικά εισιτήρια των σιδηροδρόμων. Το όνειρό μου να αγοράζω ένα, τρένο, ένα εισιτήριο τρένου στο Wigam έχοντας και να καταλήγω στη Βαρκελόνη, ίσως είναι κάτι που θα συμβεί, θα συμβεί ε, τη, στη διάρκεια της ζωής μου. Ελπίζω να τα καταφέρετε, να με ικανοποιήσετε. Χαιρετίζω επίσης ε, το θέμα της ε, κοινωνικής ατζέντα για τους ναυτικούς. Είναι κάτι που είχε καθιστορήσει πολύ και είναι πολύ καλό ότι ασχολείστε πλέον με αυτό. Για τις υπηρεσίες δάφους στα αεροδρόμια. Ένα αεροδρόμιο μου είπε ότι δεν θέλουν ανταγωνισμό. Άλλα αεροδρόμια μου λένε ότι υπάρχει υπερβολικός ανταγωνισμός σε αυτόν τον τομέα. Και αν σας πω τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια στην Ευρώπη δίνουν μια τελείως εκ διαμέτρου αντίθετη ε, απάντηση, Ίσως χρειαστεί να αυξήσουμε τον, αριθμό, τον, τον ελάχιστο αριθμό των ατόμων από 2 3 ε, σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες εδάφου στη Φραγκφούρτη και να περιορίσουμε και να προβλέψουμε ένα μέγιστο αριθμό για να βοηθήσουμε ε, ένα αεροδρόμιο όπως το Heathrow που έχει 27 ground handlers και εξακολουθεί να έχει προβλήματα. Θα ήθελα, με ενδιαφέρει λοιπόν πάρα πολύ να δω τι θα προτείνετε. Για τον ενιαίο ουρανό, ξέρω ότι ανησυχεί για αυτό το θέμα ο κλάδος. Χθες μου το είπανε σαφέστατα αυτό. Υπάρχει νομική υποχρέωση από πλευράς κρατών μελών και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη ανταποκρίνονται στις νομικές τους υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Ο κύριος ε, Τζασμπόσκι ασχολείται με αυτό το θέμα. Εγώ όταν ο κύριος Γεζεμπόφκη συναντήσει τους Γερμανούς και Γάλλους υπουργούς ε, ε, θα ήθελα να είμαι παρόν, διότι θα είναι πιστεύω μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση να παρακολουθήσει κανείς αλλά είναι γεγονός ότι πρέπει να δώσουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να μου πείτε λίγα πράγματα για τις τελευταίες εξελίξεις ό,τι αφορά την ασφάλεια των αεροπορικών εμπορευματομεταφορών. Μας μιλήσατε για ασφάλεια, αλλά τι ακριβώς θέλετε να προτείνετε εδώ. Στην προηγούμενη συζήτηση είχα πει Μιλάμε για όλη την αλυσίδα της, στον τομέα της αεροπορίας, με εμπορεύματα, για τη μεταφορά εμπορευμάτων για όλη την αλυσίδα, μιλάμε μόνο για τα αεροδρόμια. Αν μιλάμε μόνο για το αεροδρόμιο αυτή είναι η τελευταία γραμμή άμυνα, όπως είπα προηγουμένως. Αν αρχίσουν να περνάνε, να ξεφεύγουν ε, ορισμένα αντικείμενα, θα πρέπει να ξαναδούμε σε βάθος το θέμα της ασφάλειας και νομίζω ότι μου μείναν ακόμα πέντε δευτερόλεπτα από τα δύο λεπτά που είχα βάλει δώσει στον εαυτό μου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα αφήσω το θέμα των εμπορευμάτων και της ασφάλειας. Θα επανέλθω στο θέμα των εμπορευμάτων και της ασφάλειας γιατί, ε, ε, το, ε, για το τέλος, γιατί τέθηκε από άλλους ομιλητές. Για τα υπεροκιάνια δεν ε, έχουμε ακόμα καταλήξει οπουδήποτε. διερευνούμε διάφορες, τις διάφορες πτυχές ε, του θέματος. Δεν υπάρχει ακόμα τίποτα το συγκεκριμένο. Για το χρονοδιάγραμμα, δεν κατάλαβα ακριβώς ε, τι θέλετε. Το χρονοδιάγραμμα του, του φόρτου εργασίας το έχω εδώ. Ιούλιος 2011 για το χρονοδιάγραμμα θα έχουμε το, τις κατευθυντήριες γραμμές για τα τεντή και μετά εκεί θα αρχίσουν τα, τα, σοβαρά θέματα θα πρέπει να καθορίσουμε τις προτεραιότητες για τα μεγάλα έργα και θα έχουμε στο δεύτερο ήμιση του 2011 σοβαρές συζητήσεις ώστε όλα να είναι έτοιμα πριν από το 2014. Αυτή λοιπόν θα είναι η περίοδος για αυτές τις πολύ δύσκολες συζητήσεις. Το Σεζάρ, για, το, Σεζάρ όλα προχωράνε κατευχήν. Έχουν ληφθεί αποφάσεις και προχωράει η ανάπτυξη του προγράμματος. Το θέμα είναι η υλοποίησή του. Ο κύριος Ζεζεμπόφσκι συναντήσε τους δύο υπουργούς ήδη και επέζησαν οι δύο υπουργοί από αυτή τη συνάντηση. Ρωτάει ο πρόεδρος αντιλαμβάνεστε ότι απο... Ε, οσμίζεται κανείς ότι υπάρχουν, υπάρχουν κάποια προβλήματα. Βεβαίως μιλάμε για ένα σημαντικό πρόγραμμα, έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες, είναι η καλύτερη λύση, καλύτερη τεχνική λύση στον κόσμο αυτή τη στιγμή το ΣΕΖΑΡ. Εάν δεν το εφαρμόσουμε εμείς, κάποιοι άλλοι θα το εφαρμόσουν, οι Ινδοί ή οι Αμερικάνοι οπωσδήποτε. για διαφορετική χρέωση των ε, πιστοτικών καρτών για την αγορά εισιτηρίου. Αυτό δεν είναι κάτι που το έχω ακούσει. Βεβαίως δεν εμπίπτει στη δική μας αρμοδιότητα. Στις ακροάσεις διαπίστωσα ότι τα, οι άνθρωποι έχουν, έχουν πραγματικά αγανακτήσει με την υπερβολική συμφόρηση, τα μποτιλιαρίσματα. Ε, στις μεταφορές. Αν μπορούμε λοιπόν να δοκιμάσουμε, να προωθήσουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για έξυπνες πόλεις, για έξυπνες μεταφορές με πίνακα βαθμολόγησης και όλα τα σχετικά και το ίδιο ισχύει για την οδική ασφάλεια. Το πρόγραμμα λειτουργεί αποτελεσματικά. Μπορεί να μην πέτυχε απόλυτα τους στόχους τους, αλλά είχαμε μια μείωση άνω του 40% των τροχαίων ατυχημάτων και δεν μιλάμε για νομοθετικό κείμενο, μιλάμε για ένα κείμενο που κινητοποιεί όλη την κοινή γνώμη και την ευαισθητοποιεί στα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι κάτι που μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να το κάνουμε και για τις αστικές μεταφορές. Το θέμα των εισιτηρίων, των ηλεκτρονικών εισιτηρίων θα το δείτε να συμβαίνει, διότι υπάρχει μεγάλη δέσμευση για την εφαρμογή του από τη Γαλλία και την Ισπανία. Και προς ορισμένες κατευθύνσεις υπάρχει ήδη αυτή η δυνατότητα. Όχι, δεν μπορείτε να αγοράσετε από τους βελγικούς σιδηροδρόμους ένα εισιτήριο για να πάτε στη Γερμανία. Αλλά θα το δούμε το θέμα, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες, υπάρχουν ε, πολλά κεκτημένα συμφέροντα, πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να ρυθμιστούν, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε θετικές εξελίξεις. Η κοινωνική ατζέντα για τους ναυτικούς θα συζητηθεί του χρόνου, οπότε θα προταθεί και μία δέσμη μέτρων, συνάντηση εκπροσώπους των συνδικάτων του κλάδου για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί μιλάμε για σφαιρικό παγκόσμιο θέμα. Η οι ώρες ανάπαυσης των ε, οδηγών είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έγινε τίποτε. Ο χρόνος οδήγησης, μέσα στο χρόνο οδήγησης, περιλαμβάνεται και μία περίοδος ανάπαυσης. Κάτι που εφαρμόζεται καλύτερα ή χειρότερα ανάλογα με τις χώρες. Αλλά είναι κάτι που, έχει, που προβλέπεται ήδη και αν έχετε συγκεκριμένες προτάσεις δώστε μου τες διότι θα μπορέσω κάτι να κάνω. Ο χρόνος οδήγησης είναι θέμα ασφάλειας και μπορούμε ε, εκεί κάτι να κάνουμε. Κάποια παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο. Μα είναι ό,τι προβλέπει η νομοθεσία το εφαρμόζουμε. Δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν έχει γίνει τίποτε. Υπάρχουν διαφορές από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, σε ό,τι αλλά, η οδηγία, ε, του... αλλά αυτά που προβλέπει η οδηγία εφαρμόζονται. Ασφάλεια και προστασία στην αεροπορία. Η αεροπορία είναι πολύ ευαίσθητος τομέας, οπωσδήποτε Γι' αυτό όλοι πρέπει να περάσουν από ελέγχους ασφάλειας. Αν θέλετε να πετάξετε πρέπει να περάσετε από τον έλεγχο. Αυτό είναι απαράβατος κανόνα γιατί για να σώσουμε, να σώσουμε ζωές είναι μεγάλη προτεραιότητα. Για τα ε, σαρωτές μια εξέλιξη της τεχνολογία. που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όσο περισσότερο αναπτύσσεται αυτή η τεχνολογία θα είναι η καλύτερη και η πιο άνετη λύση. Δεν χρειάζεται να έχουμε διάφορες βαθμίδες ασφάλειας, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα ε, για το οποίο ε, έχετε ήδη μιλήσει. Οι οδικές εμπορευματοφορές. Το βασικό μου μήνυμα προς την κοινή γνώμη είναι κάτι που θα το επαναλάβω. Για τη ε, ασφάλεια των, ε, της μεταφοράς, αεροπορικής μεταφοράς εμπορευμάτων είναι κάτι το πολύ σημαντικό που ελέγχεται από τις εταιρείες, που ελέγχεται από τα αεροδρόμια υπάρχουν ειδικοί μεταφοροί, υπάρχουν ορισμένοι, μετα... υπάρχουν... όλοι οι μεταφορείς ελέγχονται, όλοι οι μεταφορείς τους οποίους παραδίδεται ένα δέμα ελέγχονται. Το σημαντικό δεν είναι οι διάφορες βαθμίδες ελέγχου στα αεροδρόμια. Χρειάζονται γιατί είναι αποτρεπτικό στοιχείο. Αλλά βεβαίως όλα αυτά τα συστήματα δεν θα οδηγούσαν πιθενά, πουθενά αν δεν είχαμε τη δυνατότητα να συγκεντρώνουμε πληροφορίες που μας λένε πού πρέπει να εστιάσουμε τους ελέγχους ασφαλείας. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε ότι δεν πρέπει να μεταφέρονται had to be done before. Uh, στα αεροπλάνα. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Αν θέλει κανείς να χρησιμοποιήσει το αεροπλάνο, πρέπει να έχει υπόψη του και να έχει επίγνωση του γεγονότος ότι να αναλαμβάνει κάποιους κινδύνους. Η ιδέα που προτάθηκε χθε ήταν να υπάρχει μία μαύρη λίστα αεροδρομίων. Είναι κάτι που μέχρι τώρα έχει απορριφθεί. Αλλά για σκεφτείτε το. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια μαύρη λίστα αεροδρομίων αλλά μπορούμε να πούμε ότι το αεροδρόμιο των Βρυξελών ή το Χίθρου είναι τελείως απαλλαγμένα από τον κίνδυνο καθόλου, διότι οι τρομοκράτες είναι πάρα πολύ έξυπνοι ή μπορούμε να δώσουμε ένα πιστοποιητικό στις μεγάλες εταιρείες διοικητικής μέρημνας και στις μεγάλες εταιρείες μεταφορών που είναι πολύ υπεύθυνε και ελέγχουν τα πάντα, όχι. Πιστοποιητικό ότι είναι απόλυτα ασφαλής δηλαδή μπορούμε ίσως να δώσουμε πιστοποιητικό σε κάποιες εταιρείες τις οποίες έχουμε πιο πολύ εμπιστοσύνη. Τότε ένας τρομοκράτης με τρομοκρατική οργάνωση θα μπορέσει να ε, δημιουργήσει μια εταιρεία η οποία θα πάρει αυτό το πιστοποιητικό σε δύο χρόνια. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε εμπιστοσύνη στις εταιρείε και στα αεροδρόμια που λειτουργούν αποτελεσματικά, αλλά και αυτές και αυτά πρέπει να υπόκεινται σε περιοδικούς ελέγχους. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει απόλυτος έλεγχος ε, των πάντων, διότι δεν έχουμε τα μέσα για να το κάνουμε αυτό. Αν πιστεύετε ότι μπορούμε να έχουμε άτομα και μηχανήματα που θα μας εξασφαλίσουν απόλυτη ασφάλεια, αυτό είναι κάτι που δεν ισχύει. Πρέπει τα μέτρα ασφαλείας μας να στηρίζονται στην εμπιστοσύνη και όχι στη δυσπιστία, διότι μόνο τότε θα εντοπίσουμε συγκεκριμένους κινδύνους, διότι επαναλαμβάνω, κίνδυνοι υπάρχουν πάντα. Δεν υπάρχει μηδενικός κίνδυνος, αλλά μπορούμε τον κίνδυνο να τον περιορίσουμε και να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στην καταπολέμηση και στην εξουδετέρωση των κινδύνων που υπάρχουν. Χθε διατυπώθηκαν ορισμένες προτάσεις από τους υπουργού εσωτερικών που συνεδρίασαν ε, και είπαν, είπαν ότι πρέπει και συζήτησαν τη δυνατότητα να, αλλάξουν, να αλλάξει ριζικά το σύστημα. Πώς θα γίνει κάτι τέτοιο και θα ε, ε, επιφέρει αλλαγές ε, ουσιαστικές και χρήσιμες μια τέτοια προσπάθεια. Την περασμένη Παρασκευή είχαμε μια συνεδρία εμπειρογνωμόνων που ήταν πολύ χρήσιμη και η οποία συζήτησε πώς, πώς πρέπει να αντιδράσουμε τώρα αντιμετωπίζοντας ε, τις, ε, τωρινές, τις σημερινές απειλές. Σας ευχαριστούμε πολύ, Επίτροπε, για την ε, συνεισφορά σας σήμερα το πρωί και επειδή απαντήσατε στις ερωτήσεις των μελών, προσβλέπουμε στη μελλοντική μας συνεργασία και για του χρόνου Βλέπετε ότι είμαστε, παρουσιάζουμε μεγάλο, δείχνουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Πολλοί δεν ξέρουν γιατί μιλάνε. Βάση περιπτώσει, αστείευομαι. Θα συνεργαστούμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.